Καλημέρα και καθίστε παρακαλώ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι για να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι στη δεύτερη αυτή ημέρα της ε, συνεδρίασης της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 12.30 σήμερα και έχω μια ανακοίνωση. Χθες οι συντονιστές απεφάσισαν να διεξαχθεί διάσκεψη ακρόαση μάλλον στις 9 Φεβρουαρίου για τα θέματα της Ουγγαρίας εφόσον βέβαια εγκριθεί η ακρόαση από το Προεδρείο. Εάν δεν προβληθούν ενστάσεις η πρόταση θα θεωρείται εγκεκριμένη από την Επιτροπή Θεμελιδών Ελευθεριών. Και ας έρθουμε τώρα στην σημερινή μας ημερήσια διάταξη, όπου στο υπαριθμό 21 θέμα το πρώτο θέμα θα είναι η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως του συναδέλφου μας κ. Παπα-Νικολάου για τις τεχνικές τροπολογίες που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κώδικα συνόρων Σέγγεν. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον ε, εισηγητή και μετά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τα πρώτα σχόλια και μετά θα δώσω το λόγο στην αίθουσα. Κύριε Παπα-Νικολάου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σήμερα η συζήτησή μας στρέφεται γύρω από τεχνική τροπολογία του δεύτερου κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Από τότε που εγκρίθηκε το 2006 ο σχετικός κανονισμός υπήρξαν εξελίξεις και στο νομικό αλλά και στην πρακτική εφαρμογή. Εγκρίθηκε και ο κανονισμός για τις προξενικές θεωρήσεις, καθώς και τα σχετικά συστήματα και βέβαια εγκρίθηκε και ο κανονισμός Frontex, λαμβάνοντας αυτά υπόψη και, με, και εν ώψη των πρακτικών εμπειριών των χωρών μελών από την εφαρμογή του κώδικα συνόρων Σέγγεν, είναι ορθό και συμφωνούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει τον κανονισμό για το δεύτερο κώδικα συνόρων για να τον ευθυγραμμίσει με τις εξελίξεις ε, πρακτικές και νομικές στο επίπεδο της Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές του θέματος για τη συνεργασία τους στην πρώτη φάση τις κυρίες Μπόσκουρτ, Βέμπερ, Σντανόκα, Έστρατ και Κίρκοπ και κύριο Κίρκοπ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ και την Helen Κάλες και το επιτελείο της, της γραμματείας δηλαδή της Επιτροπής ΛΥΜΕ για την υποστήριξή τους. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία με την οποία είχα θαυμάσει επικοινωνία και ελπίζω η επικοινωνία αυτή να συνεχιστεί και με τη Δανέζικη Προεδρία. Δεν πρόκειται για συζήτηση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εισαγωγή μεθοριακών ελέγχων, δηλαδή η τροποποίηση του άρθρου 23. Δεν πρόκειται λοιπόν γι' αυτό, ούτε ε, συζητούμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για, τις, για τους ευφυείς ελέγχους των συνόρων. Νομίζω ότι οι κύριοι Βέμπερ και Κοέλιο θα έχουν κάποιες δυσκολίες σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 23. Αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Πρόκειται για τεχνική έκθεση και εφαρμόζεται σε όσους περνούν τα σύνορα και αναφέρεται στα πρότυπα των σύνορων. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες των τροπολογιών, θα ήθελα μάλλον να τονίσω ορισμένα ε, που θα ήθελα να ακούσω τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πρώτα, Κομισιόν και Συμβούλιο συζήτησαν διαμακρών για τον καλύτερο δυνατό υπολογισμό τη διάρκεια, τη διάρκεια ενό ενός πρόσωπου θα επιθυμεί να παραμείνει στην επικράτεια μια χώρα μέλου. Και τώρα που το συζητούμε και παρόλο που έχουμε τι σχετικέ διατάξει στον δεύτερο κώδικα συνόρων, σε πολλέ χώρε μέλη εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα υπολογισμού. Και έχουμε και πολλά σχετικά παραδείγματα. Γι' αυτό το λόγο και πάλι γίνεται προσπάθεια από τα δύο άλλα θεσμικά όργανα και από εμά βέβαια να γίνει το σύστημα πιο εύχριστο και να συνδυάζει μια προσπάθεια επίλυση όλων των αναγκών και βέβαια να είναι και τεχνικά υποστηρίξιμο. Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη νέα πρόταση, μπορεί όντω να αποβεί αποτελεσματική. Θα διευκρινίσω πρώτα ότι προτείνουμε να υπολογίζεται ο, ο χρόνος σε ημέρες και όχι σε μήνες, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποίησεις μεταξύ χωρών μελών που ε, προκύπτει πρόβλημα αν είναι 30 ή 31 ημερών ο μήνας. Δεύτερο, πρέπει να θεωρηθεί ως κινητό πλαίσιο χρόνου. Αν δηλαδή κάποιος εισέλθει στη, την 1η Ιουλίου στην επικράτεια μιας χώρας μέλους, πηγαίνουμε πίσω 180 ημέρε για να δούμε εάν έχει μείνει μια περίοδο μέχρι 90 ημερών, αν για παράδειγμα οποιαδήποτε μέρα μετά από αυτές κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το νόημα του κινητού χρονικού πλαισίου. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν γνωρίζουμε πόσες μέρες έχει παραμείνει τις τελευταίες 180 ημέρες και έτσι γνωρίζουμε πόσες μένουν υπόλοιπες. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διευκρινήσεις που έχει επιφέρει την τελευταία περίοδο. Τα δε έγγραφα που μου διαβίβασαν και για αυτά την ευχαριστώ δηλαδή. Ευχαριστώ επίσης τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, κ. Φάμπιαν Λούτς, για την τροπολογία 14 το κάναμε με αυτή την ε, ε, έννοια ώστε να είναι εύχριστο και να μην μπερδεύεται κανένας. Δεύτερο, στη διάρκεια της σύνταξης του εγγράφου λάβαμε υπόψη και θέματα θεμελιδών ελευθεριών και δικαιωμάτων όπου αυτό ήταν δυνατόν, κυρίως για ανηλίκους και αναπήρους, τροπολογίες 16, 27 και 28. Και ιδιαίτερα στην 17 προσπαθούμε να αναρμονίσουμε τον κανονισμό με τις ήδη εγκριθεί οδηγίες για να υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ του κειμένου και των δικαιωμάτων των ατόμων να λαμβάνουν ε, πληροφορίες γραπτές ή με άλλους τρόπους. Και επίσης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται χώρες μέλη να μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερη ρύθμιση για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται μέσα στην Ισέν. Γι' αυτό δηλαδή ε, η ηθική λωρίδα λοιπόν, αλλά εδώ τα πράγματα <clears throat> μπορούν να είναι λίγο, μπορεί να προκαλέσουν λίγο σύγχυση. Κάποιο ο οποίο δεν καταλαβαίνει καλά αγγλικά ενδέχεται να μπερδευτεί, να πάει δηλαδή στη λωρίδα αυτή για να λάβει την προξενική θεώρηση ή να πάει εκεί όπου δεν υπάρχει προξενική θεώρηση και ξέρω ότι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προσπάθησαν να βρουν άλλες λύσεις. Εμείς προτείνουμε σήμερα μια λύση. Προτείνουμε λοιπόν να αλλάξουμε τη διατύπωση να λέει visa not required. Δεν απαιτείται θεώρηση. Διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι σαφέστερο και δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνιών από τους ε, ε ταξιδιώτες. Αναφέρομαι στις 18 και 19. Συμφωνούμε επίσης με Κομισιόν και Συμβούλιο ότι θα πρέπει αντί ε, joint να είναι shared crossing points με κοινή δηλαδή ευθύνη για τον έλεγχο των συνόρων αυτών μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών. Η Επιτροπή προτείνει πιο αναλυτική λίστα των ε, ε, ρητρών προφύλαξης για την εφαρμογή τους. Η Πολωνική Προεδρία ήθελε μια πιο εύκαμπτη ε, διάταξη. Έχουμε λοιπόν από τη μια την Επιτροπή που περιγράφει όλες τις ευθύνες που θα περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή, σύμφωνα βέβαια και με το κοινοτικό κεκτημένο και από την άλλη μεριά το Συμβούλιο λέει πρέπει να συμφωνήσουμε και να σεβαστούμε όλα αυτά, αλλά στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμόζεται τόσο αναλυτική διάταξη. Με τη δική μας έκθεση και τη δική μας πρόταση εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές προτάσεις που θα επιτρέψουν χώρε μέλη να έχουν κάποια ευκαμψία για να κάνουν διμερεί συμφωνίες από τη μια, αλλά θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασκεί τις αρμοδιότητές της, να εξετάζει τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο και να δίνει την τελική έγκριση. Στην πρότασή μας λοιπόν προσφέρουμε περιθώριο στις χώρες μέλη για να ε, διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες και από την άλλη μεριά διασφαλίζουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία, ο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όλων των σχετικών διατάξεων αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια, α διευκρινίσω επίση ότι περιλαμβάνουμε και μια διάταξη, ευχαριστώ την κυρία Βέμπερ για ε, την προσπάθεια αυτή ιδίω, που λέει ότι η χρήση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται να γίνεται, να διαβιβάζεται δηλαδή σε συνοριακούς φρουρού άλλων τρίτων χωρών. Ορισμένοι θα πούνε ότι αυτό είναι υποθετική περίπτωση. Αλλά έχουμε ήδη περιπτώσεις όπως είδαμε και στη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας ή Ουγγαρία και Κροατίας. Πράγματι τέτοιε συμφωνίες, εάν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της, του χώρου Σέγγεν. Έρχομαι και στην ε, τροπολογία 30 σχετικά με τις δυνατότητες χωρών μελών να ζητήσουν από υπηκόους τρίτων χωρών να παρουσιάζονται όταν, όταν εμφανίζονται σε επικράτειες, τρίτων, ε, χωρών μελών. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διαγραφή, κατάργησή της. Ωστόσο είναι λογικό, διότι ορισμένες χώρες μέλη θέλουν να την κρατήσουν ακόμη και γι' αυτό προτείνουμε εμείς να περιληφθεί στο κείμενο ως δυνατότητα αλλά όχι ως υποχρέωση. και να επαφιέται στη διακριτική ευχαίρεια των χωρών μελών, όπω είπα, δυνητικά. Τέλο, ορισμένε τροπολογίε έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, όπω η 26, η οποία δίνει μεγαλύτερο περιθώριο στην εποπτεία των συνόρων, καθώ και άλλε όπω η 32 που δίνουν τη δυνατότητα χρήση περισσότερων στατιστικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση τη εφαρμογή του κώδικα συνόρων Σέγγεν και μερικέ ακόμα τεχνικέ τροπολογίε που βελτιώνουν το κείμενο Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ε, τροπολογία 9 με δύο νέους ορισμούς για τη διάβαση των συνόρων και 10 των υπεράκτιων εργαζόμενων. Ελπίζω να μην ειμαι Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπα-Νικολάου. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Λούντ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. να επισημάνω ότι παρότι είναι μια τεχνικού χαρακτήρα πρόταση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίσονο σημασία. Στο αντίθετο, στην πρακτική καθημερινή ε, πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ταξιδιώτες και συνοριοφύλακες, αυτή η πρόταση είναι πολύ σημαντική. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει την επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων και να μειωθεί ε, η περιττή γραφειοκρατία θα διευκολύνει λοιπόν την καθημερινότητα των συνοροφυλάκων και των επιβατών. Θυμηθείτε πόσο ε, μακρές είναι οι ουρές αναμονής. Και επίσης θα μας δώσει και οικονομίες κλίμακας. Αυτή τη στιγμή μιλώ για τους προτινόμενους κανόνες για τα κοινά συνοριακά περάσματα. Σε ό,τι αφορά Επίσης, το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αυτόν τον τρόπο, με αυτό που προτείνουμε, θα ενισχύσουν περαιτέρω τα δικαιώματα αυτά. Να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι η Επιτροπή και η Κρότες όψεω συμφωνεί με την συντριπτική λιοψηφία των προτινόμενων τροπολογιών. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε μεγάλο βαθμό οι τροπολογίε είναι και έχουν ως γνώμονα να βοηθήσουν την πρακτική άσκηση του ελέγχου στα σύνορα. Ένα μόνο σχόλιο, κάτι που επισημάναμε και στο Συμβούλιο όταν παρουσιάσαμε την πρότασή μας. Η πρόταση αυτή είναι τεχνική με πάρα πολλά θέματα, αγκαλιάζει πολλά θέματα προτείνουμε 20 τροποποιήσεις σε 20 διαφορετικά άρθρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να περιορίσουμε τις τροπολογίες και να μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Ο κίνδυνος που ελοχεύει και στο Συμβούλιο είναι ότι τα κράτη-μέλη με τις ε, προτάσεις τους, θεμητές σε μεγάλο βαθμό, ανοίγουν πάρα πολύ τη συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την προσοχή μας στις προτινόμενες αυτές αλλαγές, ιδάλλως δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. Θα ενθάρρυνα λοιπόν όλους να έχουν μια κάποια αυτοπιθαρχία στη συζήτηση και να εστιάσουν στις προτάσεις τροποποίησης που κάνουμε εμείς. Στο μέλλον, έχοντας λάβει υπόψη αυτή τη συζήτηση τώρα, θα κάνουμε και νέες προτάσεις. Για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την πρόταση σύντομα, είναι καλό να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δικές μας τροποποίησεις. Και ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή γιατί σε μεγάλο βαθμό κράτησε αυτήν την αυτοπιθαρχία. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε περαιτέρω καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Λούτς. Εξ ονόματος της Προεδρίας, ο κύριος Χόλμαν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Η Προεδρία θα ήθελα να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίε επί τη πρόταση αυτή τη Νομόδια Ομάδα Εργασία του Συμβουλίου. Στόχο Προεδρία είναι να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή πριν τα τέλη τη Προεδρία μα. Η Προεδρία είναι πεπισμένη ότι αυτό είναι εφικτό. Περιμένουμε βεβαίω να δούμε τι τροπολογίε που θα υποβληθούν στο σχέδιο τη έκθεση του κ. Παπα-Νικολάου. Όπως είπε και η Κομισιόν, η Προεδρία προσπάθησε να περιορίσει τη συζήτηση στα θέματα που έθεσε στην αρχική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η τροποποίηση του κώδικα των να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί ταχύτερα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα για το Συμβούλιο, όπως επεσήμανε ο κύριος Παπα-Νικολάου, είναι η απλοποίηση του υπολογισμού της συγκεκριμένη περίοδου παραμονής στον χώρο Σέγγεν για τους προς δηλαδή των ταξιδιωτών. Υπάρχει μια γενική συμφωνία στο Συμβούλιο ότι οι αλλαγές στο άρθρο 5.1 για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής θα πρέπει να ισχύει για τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από θεώρηση, αλλά και σε υπηκόους τρίτης χώρας για τους οποίους απαιτείται θεώρηση. Για το λόγο αυτό θα ήταν αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κώδικας θεωρήσεων σύμφωνα με, το νέο κείμενο στο άρθρο 5 όπως και σχετικές άλλες διατάξεις ε, των σχετικών νομοθετικών πράξεων που αφορούν στις θεωρήσεις. Για τα υπόλοιπα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου για την καλή συνεργασία που είχαμε και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώ αυτό το φάκελο ε, του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Παπα-Νικολάου, για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Πράγματι, προτεραιότητα είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο χώρο Σέγγεν. Τροπολογία 2. Η ευθύνη για την ε, διαχείριση των κοινών εξωτερικών σύνορων Σέγγεν στα πλαίσια της αλληλεγγύης και του ίσης κατανομής των βαρών και έναν αποτελεσματικό έλεγχο των σύνορων. Τροπολογία 6. Η πλειοψηφία τροπολογιών μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών, όμως έχουμε κάποια προβλήματα με τροπολογία 30, που προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προβλέψουν νομικά υποχρέωση για επικούς της χώρας να αναφέρουν την παρουσία του στην επικράτεια και επικράτεια του μέλους. Αυτό το μέτρο ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε ε, από κράτος μέλος και διαγράφει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ήταν, ήταν καλό και θα εκτιμούσαμε να παραμείνει εκτός της πρότασης. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Σβέμπα. Thank you very much. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλοι επιμένουν από ό,τι βλέπω ότι η έκθεση αυτή είναι τεχνικής φύσεως. Συχνά όμως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ό,τι είναι πολύ τεχνικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ σημαντικό. Μέσα, αυτό, μέσα από τεχνικά, αν θέλετε, στοιχεία, θέλουμε με να προσθέσουμε τα συμφέροντα των μελών, αλλά ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των προσώπων, των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Επικρατεία. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα. Εργάστηκε πολύ καλά μαζί μα, με όλου του κοιόδη και βλέπετε τελικά ένα σχέδιο έκθεσης που ακολουθεί μια σοφή προσέγγιση καθώς έλαβε υπόψη αυτά που είπαμε στις κοινέ συνεδριάσεις ή και διμερώς. Υπ' αυτή την έννοια ε, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου και την ευχαρίστησή μου για αυτή τη συνεργασία που είχαμε. Η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει μια ισορροπημένη προσέγγιση, προστασία δηλαδή και των συμφεροτοκράτων μελών, αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, προσώπων. Αν τώρα θεωρηθεί αναγκαίο να γίνουν κάποιες άλλες τροπολογίες για καλύτερη διασαφήνιση κάποιων όρων, αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε συνεργασία, σε μια κοινή προσπάθεια. Κατανοώ βεβαίω και τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν όμως κάποιες φήμες ναι, εντάξει, μπορεί να σε κλείσουν κάποια στοιχεία στην έκθεση, αλλά πιστεύω ότι αν κάνουμε μια κοινή προσπάθεια θα καταλήξουμε σε κάτι καλό για όλους. Παρά τα αυτά θέλω να πω ότι τίνω και εγώ να συμφωνήσω με την προλαλή σας για το άρθρο, η μάλλον 30. Πιστεύω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα περαιτέρω. Πέραν τούτου θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή. Ε, Mrs. κυρία Head. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον εισηγητή, για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Δυστυχώ δεν είχα τον χρόνο να διατρέξω όλε τι τροπολογίε. Μπορώ να θέσω ίσω ένα χαζό ερώτημα, αλλά κατάλαβα καλά. Θα αυξήσουμε την διάρκεια σε ημέρες. Δηλαδή, πάμε στις 30 ημέρες, αλλά θα αλλάξουμε τον αριθμό των ημερών. Δεν τι ακριβώς εννοούσαμε αυτόν τον μήνα που αναφέρατε πριν. Ευχαριστώ. Εντάξει. Θα επαναλάβω. Ίσως να κατάλαβα λάθος, αλλά θα αυξήσουμε τον αριθμό των ημερών. Αυτό είπατε. Τον αριθμό των ημερών για τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μείνουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε από τώρα ένα μήνα στις 30 ημέρες. Αλλά αυξάνεται ο αριθμό των ημερών. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Σεγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν αναφερόμαστε σε αύξηση του αριθμού των ημερών. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι 90 ημέρες υπολογίζονται, που, αυτές που υπάρχουν ήδη δηλαδή στον κώδικα. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε έναν τρόπο υπολογισμού των ημερών έξι μήνες για ένα χρόνο αν δείτε τα, κείμενα της ομάδα εργασίας των κρατών μελών, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές από χώρα σε χώρα. Επιτροπή και Συμβούλιο, λοιπόν, και εμεί συμφωνούμε, προσπαθούν να βρουν ένα κοινό τρόπο ε, υπολογισμού των ημερών, πιο, ένα πιο εύχριστο τρόπο που μπορεί να ε, είναι και τεχνικά πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό θεωρούν ότι μπορούμε να λέμε ότι για κάθε μέρα, θεώρηση, ε, μέρα που χρειάζεται θεώρηση να εξετάζουμε τις τελευταίες 100 ημέρες για να δούμε αν υπάρχουν άλλες ημέρες έως τις 90 ημέρες. Η συνολική περίοδος είναι η ίδια. Thank you for all... Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν απάντησα κατευθείαν. Μιλούσα με τον συντονιστή μου. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Έχουμε τώρα την καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επικοδομητικά με το ίδιο πνεύμα για να οριστικοποιήσουμε την ανάλυση και να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ και πάλι και είμαι στη διάθεσή σας αν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Και πάλι είναι καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίε 8 Φεβρουαρίου στι 12 το μεσημέρι και η εξέταση τροπολογιών θα γίνει στι 27 και 28 Φεβρουαρίου κατά την ε, ε, συνεδρία τη ΛΥΜΠΕ. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, 22. Και θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για την ε, πρόταση τροποποίησης ε, του κώδικα Σέγγεν της κυρία Βέμπερ. Είναι βεβαίως ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα. Η συγγήτρια κυρία Βέμπερ έχει ως στόχο να συζητήσει σήμερα μαζί μας τα κύρια στοιχεία της ε, πρόταση της Επιτροπής πριν παρουσιάσει το προσχέδιο έκθεσής της. Θα δώσω το λόγο τώρα στην συγγήτρια και μετά αν θέλει να παρέμβει η Επιτροπή, μπορεί να το κάνει και μετά θα δώσουμε το βήμα στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που λαμβάνει η χώρα συγκεκριμένα για αυτό το φάκελο, παρόλο που έχουμε συζητήσει αρκετές πτυχές που σχετίζονται με τον χώρο Σέγγεν γενικότερα, στη Λίμπε, αλλά και στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να θυμόμαστε πώς ξεκίνησα ε, όλη αυτή η υπόθεση από την πρόταση της Επιτροπής. Πέρυσι, νομίζω όλοι θυμάστε, έγινε κάτι και δεν θέλω να κάνω ε, να εκφέρω γνώμη σε πολιτικό ή νομικό επίπεδο για το τι έγινε, αλλά κάποια στιγμή η Γαλλία αποφάσισε να επανασαγάγει τους συνοριακούς ελέγχους με την Ιταλία. Εφόσον υπήρχε ένας ε, μεγάλος αριθμός ε, ε, την νησίων που είχαν φτάσει στα σύνορα τη Γαλλία και η Ιταλία έχει αποφασίσει να του δώσει θεώρηση για να ταξιδέψουν όπου θέλουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Είχαμε μια αρκετά τεταμένη ατμόσφαιρα και συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομίζω ήταν σκληρές ε, οι διαπραγματεύσεις. Όπως και να έχει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση Βέβαια το δικό μας αίτημα ήταν διαφορετικό. Το Κοινοβούλιο που πραγματικά θέλει να διατηρήσει και να βελτιώσει ό,τι μπορεί να βελτιωθεί ε, στο χώρο Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στο χώρο Σέγγεν. Το Κοινοβούλιο ήθελα, ήθελε πάρα πολύ και να το διατηρήσει αυτήν την αρχή αλλά και να τη βελτιώσει. Ζητήσαμε λοιπόν από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση. Το Συμβούλιο είχε μάλλον διαφορετική άποψη. Όπως και να έχει, η Επιτροπή κατέθεσε μια αρκετά τολμηρή και καινοτόμο πρόταση, μπορώ να πω, που προσωπικά με βρίσκει σύμφωνη, αλλά ομολογώ ότι έχει γύρει σκληρές αντιδράσεις στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα έντονες. Υπάρχει μεγάλη αντίθεση στο Συμβούλιο λοιπόν, αλλά και ένα δισταγμό, μια επιφυλακτική στάση από πλευράς Κοινοβουλίου. Ε, που φτάνει μέχρι και το βαθμό της αντίθεσης σε ό,τι αφορά τη χρήση της επιτροπολογίας. Ένα στοιχείο της πρότασης είναι ότι όταν υπάρχουν ε, ε, προβλέψιμα γεγονότα που ενδεχομένως να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη μιας χώρας, το κράτος μέλος οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή και μετά η απόφαση επανεισαγωγής ε, των συνόρων θα λαμβάνεται από την Επιτροπή μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Αυτό για τα προβλέψιμα γεγονότα. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η πρόταση Επιτροπής λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν από μόνα τους να επανασαγάγουν τους ε, μεθοριακού ελέγχου για διάστημα έω πέντε ημερών και από εκεί και πέρα θα απευθύνονται και πάλι στην Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν, ε, όπως είπα, μεγάλη αντίθεση, λέγοντας ότι το κράτος μέλος είναι αυτό που είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η δημόσια τάξη του ή ε, εθνική ασφάλεια. Αλλά και στο Κοινοβούλιο άκουσα συναδέλφου να λένε ότι η επιτροπολογία δεν είναι η κατάλληλη προσέγγιση εδώ. Εφόσον είμαι εισηγήτρια, από τότε που ανέλαβα αυτή την έκθεση, είχα αρκετές συζητήσεις με αρκετά κρατημέλη, με προεδρίες και με την Πολωνική και τώρα βεβαίως με τη Δανική, με την οποία έχω ήδη συναντηθεί πολλές φορές. Πολλές συζητήσεις βεβαίως και με την Επιτροπή. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και με τους Χιώδης ε, για να τους ενημερώσω για την κατάσταση. Πού βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. αυτή η επιφύλαξη, εντάξει, η επιφύλαξη δεν είναι πρόβλημα, η αντίθεση είναι το πρόβλημα, είναι αρκετά μεγάλη. Δύο κρατημέλη μάλιστα έχουν ε, δηλώσει ρητά, η Νορβηγία και η Ελβετία, ότι καμία απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή μέσω επιτροπολογίας μπορεί να τους δεσμεύσει ε, νομικά εφόσον δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προσπάθησα να βρω ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα κράτη-μέλη, αλλά να διαφυλάξει αυτή την ιδέα της κοινοτική προσέγγισης ε, όταν πρόκειται για επανεσαγωγή μεθοριακών ελέγχων. Και πιστεύω ότι στις περιπτώσεις αυτές των προβλέψιμων καταστάσεων. Βεβαίω τα κράτη-μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα γειτονικά κράτη-μέλη, το γειτονικό κράτος μέλος μάλλον που θα επηρεαστεί, και όταν ληφθεί η απόφαση από τα κράτη-μέλη, μένει στα κράτη-μέλη, αλλά είναι παρούσα και η Επιτροπή και το άλλο κράτος μέλος που επηρεάζεται. Ούτε η Επιτροπή, ούτε το γειτονικό κράτος μέλος έχει ε, δικαίωμα να θέσει βέτο. Γι' αυτό και πάλι αποτελεί αρμοδιότητα της, ε, του κράτους μέλους αυτή η απόφαση. Όπως και να έχει όμως, με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται αποφάσεις ε, με μια κοινοτική διάσταση. Και αυτό δίνει βεβαίως και δυνατότητα στην Επιτροπή να αιτιολογεί και να τεκμηριώσει με καλύτερο τρόπο ε, την, ε, την απόφαση της ε, εάν χρειαστεί, εάν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του κράτους μέλους. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι και η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει τις κατευθυντήρες γραμμές που όλοι περιμένουμε για να δούμε τι ακριβώς συνιστά απειλή στην εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Το συζήτησα αυτό το θέμα με κάποια κρατημέλη. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό, αλλά θα δούμε. Για τις ε, έκτατες ε, περιπτώσεις, Θέλαμε να επεκτείνουμε αυτή την ε, περίοδο των πέντε ημερών κατά την οποία το κράτος μέλος να αποφασίσει μόνο του και να το πάμε στις δέκα μέρες και μετά να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα αλλά και για όλους τους κοιόδης είναι η δυνατότητα η έλλειψη αυτής να ληφθεί απόφαση όταν το μόνο πρόβλημα είναι η μετανάστευση, μεταναστευτική ροή. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά ότι ποτέ μια μεταναστευτική ροή από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί απειλή στην δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια τάξη. Γιατί εκεί η μετανάστευση είναι το πρόβλημα ε, και, και αυτό δεν μπορούμε να το υποδεχθούμε. Μπορούν να υπάρχουν και άλλε καταστάσει, όπω συμπεριφορέ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όχι η μετανάστευση αυτή καθ' αυτή. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η Γαλλία πάντα έλεγε ότι η απόφασή τη δεν ε, οφειλόταν στη μετανάστευση, στη μεταναστευτική ροή, αλλά σε ορισμένε δραστηριότητε ε, και ενέργειε που έλαβαν χώρα το ίδιο διάστημα. Υπάρχει και άλλο εξίσου σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο ιδίω, η νομική βάση. Εδώ και πάλι βλέπουμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν έχουν την ίδια γνώμη. Η Επιτροπή πρότεινε αυτή την ιδέα απόλυτα ετηλογημένη ότι η νομική βάση είναι το άρθρο 77 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο μάλλον ε, το υιοθετεί απολύτω. Το Συμβούλιο όμως λέει ότι το άρθρο 70 είναι η νομική βάση. Αυτή τη νομική βάση θέλει να χρησιμοποιήσει το Συμβούλιο. Δύσκολη καιρή λοιπόν βρίσκονται μπροστά μας. Φυσικά θα υπάρξει συντονισμό μεταξύ εμού και του κυρίου Κοέλιο, εισηγητή για την αξιολόγηση, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την νομική βάση είμαστε αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση. Η απόφαση του Συμβουλίου, την τελευταία εβδομάδα νομίζω, γνωρίζαμε την πρόθεση του Συμβουλίου, αλλά και πάλι θεωρήσαμε ότι ήταν αρκετά επιθετική στάση του Συμβουλίου απέναντι στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως είμαστε εδώ να εργαστούμε από κοινού για την νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Γιατί οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο εκπροσωπούν τους ίδιους Ευρωπαίους πολίτες που εκπροσωπούμε και εμείς. Γι' αυτό είναι δύσκολο να καταλάβω, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο κρίση, πώ είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια έλλειψη κατανόηση ε, μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και στέλνουμε πολύ άσχημο μήνυμα στου πολίτε μα και όχι μόνο σε αυτού. Εγώ ντρέπομαι όταν βλέπω ότι ε, οι ρεπουμπλικανοί ε, που κατακρίνουν τον Ομπάμα στη ΣΥΠΑ λένε ότι θα καταλήξετε σαν την Ευρώπη. Αν είναι δυνατόν Σίγουρα δεν ήταν αυτό το όραμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Ρενάτα. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά εγώ θα το πω. Καλή χρονιά, θέλω να σε ευχηθώ. Και επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια. Είχα την χαρά και την τιμή το περασμένο φθινόπωρο να παρουσιάσω στην Επιτροπή σα ε, το νέο πακέτο προτάσεων μα και χαίρομαι γιατί και εσεί κατανοείτε ότι είναι ένα πακέτο με κοινό στόχο τη βελτίωση τη ε, λειτουργία ε, του Σέγγεν και τη διακυβέρνηση Σέγγεν. Δεν ε, χρειάζεται να περιμένουμε να, να προκύψουν τα προβλήματα. Πρέπει να εξεύρουμε τρόπου ώστε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα θα λειτουργεί ομαλά. Επιτρέψτε μου να σα υπενθυμίσω τρία στοιχεία του πακέτου μα. Πρώτον, η πρόταση για την τροποποίηση του κώδικα στον Σέγγεν, και θα επανέλθω σε λίγο, η πρόταση για τον μηχανισμό αξιολόγηση Σέγγεν, εισηγητή ο κ. Κοέλιο. Και το τρίτο στοιχείο που θεωρούμε σημαντικό είναι η πρόταση βάσει της οποίας το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει δύο φορές το χρόνο να έχουν μία συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του Σέγγεν, δηλαδή για τον Ευρωπαϊκό χώρο χωρίς σύνορα. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια μιας επισκόπησης που θα έχει κάνει προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί κατά τη διάρκεια τη Ιδανική Προεδρία η πρώτη τέτοια συζήτηση θα γίνει στο Συμβούλιο τον Ιούνιο και η πρώτη επισκόπηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του Σάγκεν θα γίνει το Μάιο. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω σε μία σειρά σημείων, ιδίω αυτά που έθεσε η συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι παρότι Υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση για το μηχανισμό αξιολόγηση Σέγγεν. Αυτή είναι μια πρόταση που είναι αρμοδιό του κυρίου Κοέλιο. Πιστεύω όμω ότι δεν υπάρχει διαφωνία σε ό,τι αφορά τη νομική βάση για την τροποποίηση του κώδικα Σέγγεν. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έχει κάνει ένα ειδικό σχόλιο για την καταλληλότητα του άρθρου 26. Αυτή είναι η συζήτηση που συνεχίστηκε στην ομάδα εργασία την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η νομική βάση για την ίδια την πρόταση δεν είναι θέμα, δεν τίθεται να επιβόλει Υπάρχει πλειάδα άλλων θεμάτων που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά όχι αυτό. Επίση, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι αυτά που θα κρίνουν κατά πόσο απειλείται η εθνική του ασφάλεια και η δημόσια του τάξη. Εννοείται ότι η εθνική κυριαρχία σημαίνει ότι το κράτο μέλο αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει μια τέτοια απειλή. Και δεν είναι πρόθεση δική μα να εκδώσουμε καθεντήριε γραμμέ σχετικά με το τι αποτελεί απειλή ένατη της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι η απόφαση για το να κλείσουν ε, τα ιστορικά σύνορα είναι μια απόφαση που πρέπει να βασίζεται στην απειλή, στην δημόσια τάξη και ασφάλεια και φυσικά αυτό έχει μεγάλες συνέπειες για τις όμορες χώρες. Η πρότασή μας λοιπόν ζητά ότι το εν λόγω κράτος μέλος που αποφασίζει την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα είναι μια απόφαση αναλογική έναντι της απειλής. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτές τις αποφάσεις για την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα. Όπως πολιορθέπει η κυρία Βέμπερ, αυτό οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις στο Συμβούλιο. Αντιδράσεις που βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει κατανοητή σε βάθος η πρότασή μας. Αυτό που πολύ ορθά είπε η συγγήτρια είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τώρα ποιοι είναι οι τρόποι βάσει των οποίων μπορούμε να εγγυηθούμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχων και ισορροπιών ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία λήψη απόφαση. Βεβαίω και το κάθε κράτο μέλο είναι ο καλύτερο κριτή του τι απειλεί την εθνική τάξη και ασφάλεια. Το αναγνωρίζουμε αυτό αλλά όπω και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναγνωριστεί ταυτόχρονα και ότι υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή πώ μια επαναφορά του ελέγχου εσωτερικά σύνορα επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Έπειτα, η συγκέντρια μίλησε για την ειδική περίπτωση Νορβηγία και τη Ελβετία. Ναι, βεβαίω αυτά τα κράτη θα συμμετάσχουν στι συζητήσει για την τελική μορφή της απόφασης. Όμως, ό,τι αφορά την επίσημη διαδικασία επιτροπολογίας, αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αναγνωρίζουμε όμως όλοι πόσο σημαντικό όλες οι χώρες Σέγγεν να έχουν λόγο ε, ε, στην όλη αυτή διαδικασία που θα διαμορφώσει την τελική απόφαση. Πιστεύω λοιπόν ότι και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση αυτών των δύο χωρών. Είναι σημαντικό να έχουμε όμω μια κοινή προσέγγιση όλοι για τον επιδιωκόμενο στόχο, για τη βελτίωση αυτού του σκέλου του κώδικα των Οσέγγεν και θεωρούμε ιδίω ότι είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι αυτό το συμμερίζεται και η Δανική Προεδρία. Ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του συνολικού πακέτου για τη διακυβέρνηση Σέγγεν. Όπω είπα, οι άλλε συνιστώσει είναι η πρόταση για την οποία είναι ο κ. Κοέλιο, όπως και κάτι γενικότερο. Οι πολιτικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να δώσει το Συμβούλιο και ελπίζω εδώ να δράξει την ευκαιρία και το Κοινοβούλιο εν ώψη της πρότασης που θα υποβάλουμε το Μάιο. Ευχαριστώ πολύ. Now I the... Ας αρχίσει τώρα η συζήτηση. Ο κύριος Έντσιου πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εκτιμώ την προσπάθεια που καταβάλει η κυρία Βέβερ, που όπως συνήθως έχει προβεί σε ανάλυση σε βάθος και που νομίζω ότι η έκθεσή της θα είναι καλή. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Ιδίως διότι οι χώρες μέλη απορρίπτουν η αδίποτε διαπραγμάτευση στην βάση της Προκείμενη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι παράξενο, διότι οι χώρες μέλη και ζήτησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη δημιουργία τέτοιου κοινοτικού μηχανισμού. Ενώ τώρα κάνουν σαν να μην έχουν καμία σχέση. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο προτεραιότητες. Αφενός να προχωρήσουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και εδώ έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητες της Δανικής Προεδρίας για να συμβάλλει σε αυτό το ξεμπλοκάρισμα. Η Προεδρία έχει μια στάση ανοιχτή και επικοδομητική. Και η άρνηση συζήτησης δεν ωφελεί ούτε το Συμβούλιο, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ας μην ότι όλες μας οι δραστηριότητες οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Και η επιστροφή σε μεθοριακούς ελέγχους δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέτρο κατεξαίρεση που στοχεύει να ε, εξυπηρετήσει καταστάσεις εξαιρετικές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα. όπως είπα με εξαίρεση βέβαια όταν υπάρχουν περιπτώσεις, συνθήκες που το επιβάλλουν. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι κοινοτικό. Η απόφαση να θεσπιστούν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα δεν μπορεί να λαμβάνεται μεμονωμένα από μια χώρα μέλος. Πρέπει να είναι απόφαση που θα ληφθεί από κοινού στο επίπεδο της Ένωσης. Βέβαια, μένει το θέμα του τρόπου εφαρμογής του μηχανισμού. Το Συμβούλιο αντιτίθεται στην ιδέα αυτό να το αναλάβει μοναχά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτροπολογίας. Η Επιτροπολογία ίσως όντως να μην είναι η καλύτερη λύση και εγώ συμφωνώ. Θα πρέπει να επινοήσουμε μια διαφανέστερη μέθοδο που να εμπλέκει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ένα άλλο θεμελιώδες στοιχείο είναι ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει εντός της διαδικασίας της συναποφάσεως και για το μηχανισμό διεξαγωγής των ελέγχων και για τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σέγγεν. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Το Κοινοβούλιο δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε απόπειρα του Συμβουλίου να τροποποιήσει την νομική βάση για να μπορέσει έτσι να βασιστεί στο άρθρο 70 αντί στο 77. Το Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να απομονώσει το Κοινοβούλιο, ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ξεκάθαρα δικές μας αρμοδιότητες. Έχω πιστοσύνη ωστόσο στην Ιδανική Προεδρία. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να επιταχύνει την ψήφιση της δέσμη μέτρων για την διακυβέρνηση του Σέγγεν, διότι έχουμε ανάγκη των μέτρων αυτών για να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Ρενάτε Βέμπερ. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Ποια ωστόσο είναι τα σημαντικά στοιχεία για μας. Όπως είπε η Επίτροπος Μάλιστον χθε, ο χώρος του Σέγγεν είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μιλούμε για ελεύθερη διακίνηση και μάλιστα σε συνθήκες ασφάλειας. Το Σέγγεν δεν έχει ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε επιγόντως την δεύτερη γενεά του συστήματος πληροφοριών το SIS-2 καθώς και ένα νέο μηχανισμό αξιολόγησης για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τι θα κάνουμε όταν κάτι θα πάει στραβά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό, μηχανισμό αξιολογήσεως εντοπισμού σφαλμάτων και σωστή εφαρμογή των κανόνων του Σέγγεν. Θέλουμε όμως ευρωπαϊκό, κοινοτικό μηχανισμό. Δεν θέλουμε πια άλλα διακυβερνητικά συστήματα και δεχόμαστε μεν την ε, πανισαγωγή των μεθαριακών ελέγχων, αλλά ως ίστατο καταφύγιο, ίστατη λύση. Και θα μπορεί να, να, να επιβάλλεται σε ολόκληρο το χώρο του Σέγγεν μόνο όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που θέλετε με διαφορετικό τρόπο. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι. Το πρόβλημα, όπως είπε και η κυρία Βέμπερ σωστά, είναι ότι οι χώρες μέλη δεν έχουν ευθυγραμμιστεί και ταυτόχρονα την ώρα που η προηγούμενη Προεδρία συνομιλούσε με το Κοινοβούλιο, οι χώρες μέλη προσπαθούσαν να παραγωνίσουν το Κοινοβούλιο. Και τώρα μάλιστα συνομιλούν στο Συμβούλιο για να τροποποιήσουν την ε, νομική βάση, να πάρουν το άρθρο 70 αντί του 77, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν από τη μέση το Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος διότι η Δανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες προτιμούν το 70 αντί το 77. Δηλαδή η παρούσα Προεδρία είναι μία από τις χώρες εκείνες η οποία πρότιμα ως νομική βάση ένα άρθρο της συνθήκης το οποίο στην ουσία βγάζει απ' έξω το Κοινοβούλιο. Και όπως είπε σωστά η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, το άρθρο 70 δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να βγει απ' έξω το Κοινοβούλιο, αλλά και για να μειωθεί το επίπεδο ρύθμισης, διότι πολλές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να εγκριθούν νομίμως στα πλαίσια του άρθρου 70. Άρα θα είναι λιγότερο φιλόδοξες οι προτάσεις. Ενώ εμείς θέλουμε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ελεύθερη διακίνηση στα πλαίσια του χώρου Σένγεν. Από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν πολλά όρια αξεπέραστα. Πρώτον, ο μηχανισμό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Δεύτερο, συναπόφαση με το Κοινοβούλιο. Τρίτο, η μετανάστευση. Δεν, δεν θα θεωρήσουμε τη μετανάστευση ως απειλή, που αυτό σημαίνει η επαναφορά των μεθοριακών ελέγχων. Η έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, η πανεισαγωγή δηλαδή των ελέγχων, είδαμε για λόγους λαϊκιστικούς ορισμένες χώρες να το πράττουν και νομίζουμε ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να μπορεί να πάει επί τόπου και να, δει, να διαπιστώσει αν υπάρχει παραβίαση των κανόνων του Σέγγεν. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε την ιδέα του Συμβουλίου να επιλέξει τα χειρότερα. Για παράδειγμα, για τον μηχανισμό για τον οποίο είναι η συγκήτρια η Ρενάτε Βέμπερ, το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να παραιτηθεί όλων των υπολείπων με την εξαίρεση του άρθρου 26, που αναφέρεται στην επανεισαγωγή των μεθοριακών ελέγχων. Το Συμβούλιο δηλαδή επιθυμεί να αλλάξει τη νομική βάση από το 77 να πάει στο 70 για να διώξει το Κοινοβούλιο, δεν θέλει ευρωπαϊκό χαρακτήρα του μηχανισμού, θέλει διακυβερνητική συνεργασία και δεν θέλει να έχει καμία ε, καμία σχέση με ελεύθερη διακίνηση. Δηλαδή μόνο να βάλει τις νέες συνθήκες για την επανεισαγωγή των ελέγχων. Βεβαίω δεν βρίσκεται το ίδιο μήκο κύματο με το Κοινοβούλιο. Δεν είναι αυτό τρόπο για να ενισχυθεί το Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εκφράζω την απογοήτευσή μου. Δεν έχω απολύτω καμία ελπίδα δε ότι θα οδηγηθούμε κάπου στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και να πει ακριβώς ποια, ποια είναι η άποψή του τη προτάσει Κομισιόν και να συνεχίσει με την νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ρομέρο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι με τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Βέβε προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού εξαναγκαστική οφείλεται ουσιαστικά στην ε, μεγάλη εισρωή την Ίσιον και α, στην ε, Λαμπετούσα. Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι αυτό το προπατορικό αμάρτημα. Κοιτάξτε, σήμερα ούτε ο κύριος Σαρκόζη, ούτε ο κύριος Μόντι θα συμφωνούσαν να κάνουν αυτό που προτάθηκε τότε. Ακόμα και οι ίδιοι πιστεύω ότι σήμερα θα ήταν κατά αυτής της ε, τροποποίησης του κανονισμού. Εκείνη όμως τη στιγμή δεν χρησιμοποιήθηκε η οδηγία του 2001 για την προσωρινή άδεια που ήταν η νομική βάση εν προκειμένου. Η κατάσταση ήταν καθαρά λαϊκίστικη και καθαρά προεκλογική. Ήταν μια απόφαση καθαρά με γνώμονα τις εκλογές και για τις δύο αυτές χώρες. Και οι δύο χώρες δεν είχαν καμία εικόνα του τρόπου που θα πρέπει να αξιολογείται ο μηχανισμός Σέγγεν όπως ο κύριος Κουέλιο και τι πρέπει να κάνει κανείς σε εξαιρετικέ συνθήκες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τελικά αυτή η τροποποίηση έχει μια κάποια πηγή, φοβούμε. Καλό θα έκανε όμως η κυρία Μάλστρομ να αποσύρει αυτή την πρόταση. Είναι πραγματικά βαρβαρότητα να συγχαίει κανείς την ίδια πρόταση, τις μεταναστευτικές ροές, με, τον, ε, με τα γεγονότα και με την τρομοκρατία. Πώς γίνονταν τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή έχουμε μεγάλες πολιτικές εκδηλώσεις και απ' την άλλη έχουμε τρομοκρατική απειλή. Και για αυτούς τους δύο λόγους καταλήγουμε στην ίδια πρόταση. Α, αναγκάζει να κάτω να επαναφέρει τους ιστορικούς ελέγχου στα σύνορα. Αν μπορούμε να φανταστούμε και άλλα πράγματα και άλλους λόγους. Πώς θα τροποποιήσουμε τον κανονισμό με τόσο μη σοβαρό τρόπο. κατανοώ ότι ασκήθηκαν πιέσει στην Επίτροπο για να υποβάλει τροποποίηση στον κανονισμό. Αλλά δεν είναι σοβαρή κατάσταση. Εμεί ω Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Κατανοώ την προσπάθεια τη κυρία βέβαια, αλλά δεν είναι η χρονική στιγμή να μιλούμε για αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν και μια κοινοτική μέθοδο για να συνομιλήσουμε τα κράτη-μέλη και να δούμε ποιε είναι αυτέ οι εξαιρετικέ συνθήκε. Δεν είναι δεν είναι η στιγμή και δεν μας προσφέρει μια τέτοια κατάλληλη στιγμή αυτή η πρώτος τροποποίησης. Λογικό θα ήταν η κυρία Μάλστρομ να αποσύρει αυτή την πρόταση, να γίνει μια αξιολόγηση του συστήματος SIS και να δούμε σε ποιες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί κανείς να προβλέψει τροποποίηση του κανονισμού και να ξεκινήσουμε ένα πραγματικό διάλογο με τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή είναι στρεβλός αυτός ο διάλογος. Δεν πρόκειται να μας οδηγήσει πουθενά. Εμείς ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη θέση. Το πρόβλημα δεν είναι η νομική βάση είναι το άρθρο 70 του 77. Το πρόβλημα είναι ότι το Σέγγεν είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες, από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε για μία μεταναστευτική πίεση την νησίων που οφείλεται στην ε, εξέγερση στη χώρα τους, να οδηγηθούμε στην τροποποίηση του κανονισμού. Δεν δικαιολογείται με τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η θέση μου και να πω ότι συμμερίζομαι όλα όσα είπε ο κύριος Ένσιου και κατανόησα και την προσπάθεια της κυρίας Βεβέρ. Όμως Χαίρομαι με αυτά που ακούω από τον κύριο Κοέλιο. Ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό ώστε να αφήσουμε στην άκρη πραγματικά αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο Λόπε, κύριε Κέλλα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα υπόθηκαν και για μένα και για του πρασίνου γενικότερα η ιδέα να έχουμε μια κοινοτική προσέγγιση σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη επαναφορά των μεθοριακών ελέγχων είναι ένα πολύ λογικό σημείο. Το Σέγγεν είναι μια κοινή απόφαση, όλοι αποφάσισαν να το συνυπογράψουν και τώρα αν η Επιτροπή ζητά να γίνει κάτι τέτοιο και να τους δώσουμε μια παραπάνω εξουσία, τότε αυτό μας φαίνεται λογικό και το στηρίζουμε. Όπως είπαν όμω και άλλοι, οποιαδήποτε επαναφορά μεθοδολογικών ελέγχων θα πρέπει ε, να είναι στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Δεν, γιατί δεν αποτελεί επαρκέ ε, μέτρο για να επιλύσει προβλήματα όπως η μετανάστευση ή διαμάχες μεταξύ κρατών μελών ή εκλογικές ε, ε, μάχε ή οτιδήποτε άλλο. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, είμαι κατά της ε, έμφασης που δίνεται στην πρόταση της Επιτροπής ε, ε, στην μεταναστευτική ροή ως απειλής γιατί ενδεχομένως δεν είμαστε όλοι μετανάστες αλλά κάποιοι από εμά είμαστε. Δεν είμαστε απειλές. Δεν αποτελούμε απειλή επειδή ταξιδεύουμε μέσα στον χώρο του Σέγγεν. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, δεν είναι απειλή στην ε, εθνική ασφάλεια. Όπως και να έχει, είναι απαράδεκτο μόνο και μόνο επειδή οι μετανάστες μετακινούνται να επανεισάγονται με θεωριακή έλεγχη ε, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ακόμα και ε, μέλη της Έγγεν που δεν φροντίζουν να είναι αρκετά στεγανά τα σύνορά του και αυτό αξιολογείται από άλλους, κατά πόσο είναι στεγανά ή όχι, να, να διώχνονται από την Σέγγεν. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου την ανθρώπινη διάσταση. Συμφωνούμε με την κοινοτική προσέγγιση. Αντιτιθέμεθα με την ιδέα ότι οι μετανάστες αποτελούν απειλή και ε, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πολύ ε, ενεργό δράση όπως και στα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε κύριε Ζήπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλοι εδώ σήμερα κατανοούμε ότι πρόκειται για μια συζήτηση ιδιαίτερα ανησυχητική. Να έχουμε κατά νου τι ακριβώς οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αν έχουν προβλήματα εθνική ασφάλεια θα πρέπει να είναι σε θέση να τα επιλύουν από μόνο του. Όμω τα κράτη-μέλη αυτά που μα οδήγησαν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση δεν αναφέρουμε μόνο σε ό,τι συνέβη στη Γαλλία πρόσφατα, ούτε για την επανεισαγωγή των ε, μεθοριακών έλεγχων στη Δανία, ούτε καν για τι κάτω χώρε που ξεκίνησε και αυτή ελέγχου με τον να ε, φωτογραφίζει τα εισερχόμενα οχήματα και δεν γνωρίζουν ούτε καν οι οδηγοί για, το, για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Και σε άλλα κρατημέλη όμως βλέπουμε ότι δεν είναι σε θέση σε εσωτερικό επίπεδο να οργανώσουν τα πράγματα σωστά. Παρόλο που είχαν πει ότι θα το κάνουν. Εάν τα κρατημέλη δεν κάνουν όσα είχαν δεσμευτεί ότι θα κάνουν, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε την κοινοτική μέθοδο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν εδώ να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο ε, ε, ό,τι αφορά την αποπτία. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση με τις τρίτες χώρες για ένα σύστημα βάση αξιών. Όμως ξαφνικά τώρα βλέπουμε τους μετανάστες ως ε, απειλή. Ακούγοντα τη συζήτηση, νομίζω ότι παρά τα όσα δραματικά συμβαίνουν, θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και να εξετάσουμε το ζήτημα των προσφύγων, ε, να διασφαλίσουμε τη Σέγγεν, να, ενισχύσουμε το χώρο Σέγγεν και όχι ε, να, ε, να υπαναχωρήσουμε απέναντι στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, διαρωτώμενος γιατί η θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι τόσο διαμετρικά αντίθετες, η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να βρω είναι ότι ε, είναι θέμα νοοτροπίας. Η δική μας νοοτροπία είναι ε, η διάσταση μιας Ευρώπης χωρίς ε, σύνορα ενώ το Συμβούλιο θέλει μια Ευρώπη με σύνορα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Είναι προφανές ότι αν σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο θα οδηγηθούμε σε διαμετρικά αντίθετε ε, κατευθύνσεις. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, όχι μόνο επειδή διαφωνούμε, αλλά και επειδή κατά τη γνώμη μου, ελπίζω να κάνω λάθος, το Συμβούλιο όχι μόνο διαφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής, αλλά μάλιστα θέλει να υπαναχωρήσει στα όσα έχουμε συμφωνήσει στη Σέγγεν, διευκολύνοντας τα κράτη-μέλη να επαναφέρουν μεθοριακούς ελέγχους όποτε το επιθυμούν. Και αυτό εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο, με το δικό μας τρόπο σκέψης. Γι' αυτό και ελπίζω να εργαστούμε από κοινού σε αυτό το θέμα, να καταλήξουμε σε μια συνένεση και να είναι ανοιχτό το Συμβούλιο ε, στην ε, εξέβρεση ενός συμβασμού. Γιατί και το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό προς μια τέτοια ε, λύση. Όμως θα πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες. Ο Κάλλος Κοέλιο ανέφερε αρκετές προϋποθέσεις και εγώ έχω προϋποθέσεις να αναφέρω. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη έχουν πραγματικές εθνικ... ανησυχίες για την εθνική τους ε, ασφάλεια, ας τις συζητήσουμε βεβαίως και να κατανοήσουμε κι εμείς ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις όπου η παναφορά μεθοριακών ελέγχων μπορεί να τελογηθεί. Εξαιτίας ε, κινδύνων για την εθνική ασφάλεια. Κάνα ένα πρόβλημα εκεί λοιπόν. Συμφωνούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά, από την άλλη, υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Το δικαίωμα που έλαβαν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει ποτέ να ακυρώνονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος που δρά βάσει μιας διμερούς απόφασης ή μιας μονομερούς απόφασης μάλλον. Γιατί τότε απλώς δεν ε, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Συμφωνώ πολύ με, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένω, ότι η μετανάστευση ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρείται απειλή και κίνδυνο ε, προ την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Ακριβώ το αντίθετο θα πρέπει να ισχύει, γιατί ακόμα και αν κάποιο μπορεί να πει ότι η εθνική ασφάλεια απειλείται ε, λόγω της μεταναστευτικής ροής, τότε η επανεισαγωγή των εθνικών συνόρων αντιβαίνει στην αρχή της αλληλεγγύης. Γιατί ουσιαστικά λέμε στα κράτη-μέλη που έλαβαν ένα, δέχτηκαν ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα ότι αυτοί οι μετανάστες θα πρέπει να μείνουν εκεί, να τους κλείσουμε εκεί μέσα. Ακριβώς το αντίθετο με την αρχή της αλληλεγγύης δηλαδή μια αρχή που, στην οποία αναφερόμαστε συχνά σε αυτήν την Επιτροπή. Εγώ απευθύνω έκκληση προ την Προεδρία. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλη αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Δανική Προεδρία, ιδιαίτερα επειδή έχει μεγάλη αξιοπιστία η Δανία ε, σε ό,τι αφορά τη Σέγγεν. Γιατί ένα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν ε, πρόσφατα ήταν η άρση των ε, εμποδίων που είχε θέσει η Δανία ε, πρόσφατα. Η Δανία λοιπόν έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ κύριε Κροτσέτα. Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο έχει μια τόσο άτεγκτη στάση. Δεν είναι κατανοητό πώς σήμερα διαβάζω τον Ιταλικό τύπο, διαβάζω τη λέει η Μέρκελ. Πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική Ευρώπη. Πώς θα ενισχύσει την πολιτική Ευρώπη έτσι, με την επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει από την άλλη ότι είναι καλή και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μπροστά μας δύο εξαιρετικά ασφαλμένες προτάσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με... είναι τελικά το μόνο θεσμικό όργανο που θέλει με ριζότερο τρόπο να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη και συνεχίζει να πιστεύει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα κράτη-μέλη βεβαίως ε, ε, εκφράζονται στη στιγμή τις κυβερνήσεις τους. Το κατανοώ και αυτό. Αυτή τη στιγμή ακούμε τις φωνές των κυβερνήσεων. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το αξιολογήσω πολιτικά αυτό. Αλλά τα κράτη-μέλη εκφράζονται από συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Παρά τα αυτά και αυτές οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τους πολίτες. Και από την άλλη, εμείς θέλουμε να α, έχουμε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διαδικασία. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τη συνάδελφο την κυρία Ρομέρο. Πρέπει να θέσουμε τα πράγματα στο κατάλληλο πλαίσιο. Δηλαδή, η πρόταση αυτή γεννήθηκε σε συγκεκριμένες συγκυριακές συνθήκες. Λέει η πρόταση σε ποιε περιπτώσει θα επαναφέρουμε τον έλεγχο στα σύνορα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την επαναφορά των ελέγχων. Μα και σήμερα, μα και σήμερα δεν μπορούν να επαναφέρουν τα κράτη-μέλη των ελέγχων στα σύνορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξαιρετική περίσταση ξαφνικά αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα στα σύνορά του. Δεν έχουν το καθήκον και το δικαίωμα να προασπιστούν και την επικράτειά του αλλά και την ευρωπαϊκή επικράτεια. Βεβαίω δεν μπορούν να το κάνουν έναντι και ει βάρο άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Και εκεί είναι η ουσία. Αυτά τα σύνορα καταργήθηκαν γιατί, γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αστυνομικές και οι λοιπές διοκτικές αρχές έχουν πολλούς τρόπους να διώκουν τις ε, παράνομες, ε, αν θέλετε, δραστηριότητες και εγκληματικέ δραστηριότητες. Λέει κύριε Βέμπερ, ότι δεν μιλούμε για έλεγχο της μετανάστευσης, αλλά για τις παράπλευρες δραστηριότητες. Δηλαδή, σήμερα, αν κανείς μεταφέρει ναρκωτικά όπλα, το απαγορεύει, απαγορεύει κανείς την αστυνομία να κάνει έλεγχο σε τέτοια άτομα και μέσα στην εθνική επικράτεια. Δεν το καταλαβαίνω. Οπότε επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Ρομέρο πριν λίγο. Αυτή η πρόταση γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. 20.000 την ίση εισέβαλαν στην Ευρώπη. Ε? Και μόνο που το λέω Γελάμε όλοι. 20.000 στην ίση εισέβαλαν και πλημμύρισαν την Ευρώπη. Γελίο είναι να το λέμε. Τι κάναμε. Κάθε μέρα απευθύναμε αιτήματα για την ε, προστασία των ανθρωπικίνων δικαιωμάτων στην Ισία. Και αν τελικά κάτι επέτυχαν οι Τινήσιοι με την εξέγερσή του. ήταν γιατί υπήρχε μια θετική στάση στην Ευρώπη. Οι Τινήσιοι έλεγαν «Ζήτω η Ευρώπη, ζήτω η Ευρώπη» και μετά εμείς τους διώχναμε πίσω. Με αυτή μας τη στάση ενισχύουμε τις εθνικιστικές στάσεις, ενισχύουμε πιο ευρωκεντρική Ευρώπη που αποκλείεται από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ανάπτυξη αν δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας προς τον υπόλοιπο κόσμο, προς την νότια πλευρά Μεσογείου κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν θέλω να μιλήσω για τη Γαλλία εγώ σήμερα, γιατί θα ήταν άδικο. Κλείνω λέγοντας. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή στην Ιταλία για προεκλογικούς λόγους λέμε αστροποποιήσουμε τον κώδικα Σέγγεν. Όχι, Πρέπει ο γνώμονας μα είναι το ευρωπαϊκό μέλλον και αυτό πρέπει να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε λεπτά έχουμε ακόμη στη διαθέσή μα, λέει πρόεδρο, και τρει ακόμη συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Βέβα και θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο, αν θέλει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ να είσαστε όλοι σύντομοι. Κυρία Κιγιόν. Oui, oui, je vous Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε, πολύ, δυσ... πολύ γρήγορα, γιατί συμφωνώ και με πολλά, πολλά όσα έχουν υποθεί ήδη. Ευχαριστώ την κυρία Βέμπερ αρχικά για το έργο της. Πολλά σημεία υπάρχουν σε αυτή τη συζήτηση για τις ε, περιπτώσεις έκτατη ανάγκης, ε, για το τι πρέπει να είναι κοινοτικό ή όχι. Βεβαίως ε, θα ήθελα να ενισχύσουμε την κοινοτική διάσταση. Και εγώ νιώθω απογοητευμένη από τη στάση αρκετών κρατών μελών που θέλουν να κάνουν το Κοινοβούλιο να ε, ενδιαφέρεται κυρίως για τη μέθοδο και όχι για το περιεχόμενο, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για, τον, για ένα μηχανισμό και περί τίνο πρόκειται, για το αν κάτι είναι προβλέψιμο ή όχι. Αν κάτι είναι προβλέψιμο, έχουμε ήδη ένα μηχανισμό, δηλαδή γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε ένα επιπλέον ε, ε, στάδιο. Και αν πρόκειται για περίπτωση έκτακτη ανάγκη, γιατί μιλάμε ακριβώ για μερικέ χιλιάδε ε, άτομα που κάποια στιγμή πάνε σοριδών ε, σε ένα κράτο μέλο. Και αυτό αποτελεί πραγματική απειλή στην εθνική, σωτηρία, ε, συγγνώμη, εθνική ασφάλεια κάποιου κράτου μέλους. Και αυτό αξίζει τον κόπο να πάμε ενάντια στις αξίες της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν ε, πραγματικά να αναρωτηθούμε ποιο είναι το όφελος μιας τέτοιας ε, πρότασης για τέτοια ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Και τέλος, πράγματι πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη περισσότερο θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την γενική αξιολόγηση του Σέγγεν παρά για μια επιπρόσθετη αξιολόγηση. Κυρία Ένστ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι και εγώ σύντομη πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής. Όταν ε, έρονται η έλεγχοι στα σύνορα, αυτό είναι συμβολικό πρώτα απ' όλα και είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Τι δείχνει η άρση των σύνορων. Ότι έχουμε μια πολιτική ολοκλήρωση ε, ο χώρο Σέγγεν είναι ένα ευρωπαϊκό επίτευγμα που δεν μπορεί κανεί να το επικαλεστεί και σε πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Όταν λοιπόν μιλούμε για τροποποίηση αυτού του επιτεύγματο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν θέλουμε να κάνουμε τροποποίησεις, θα πρέπει βεβαίω να έχουμε υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις, επίγου καταστάσει και τι δικαιολογεί μια τροποποίηση του συστήματο εν γέννη. Θα είμαι ε, πολύ σύντομη. Θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. για τη μετανάστευση. Η μετανάστευση δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπήρχε εδώ και αιώνες, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα φρούριο γύρω από την Ευρώπη. Δεν μπορεί το αποτέλεσμα της πολιτικής μας να είναι να οχυρώσουμε την Ευρώπη και να την αποκλείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Θα είμαι σύντομος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η πρόταση. Στα τέλη Απριλίου υπήρξε μία διαφωνία, ένας τσακωμός, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Γαλλία και την Ιταλία για κάποιους μετανάστες από τη Βορραφρική. Αν δεν υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στι σχέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα συνεχώ. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και όταν μιλούμε για προσωρινή επαναφορά στον έλεγχο στο σύνορα, αυτό μπορούμε να το δεχτούμε και μπορεί να βασιστεί στην αμοιβή επιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Φυσικά και υπάρχουν εξαιρετικέ περιπτώσει για τι οποίε αυτό δικαιολογείται, αλλά από εκεί πέρα το Σέγγεν είναι ένα μεγάλο επίτευγμα του πολιτισμού μα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ε, συζητούμε την τροποποίησή του. Θα πιέσουμε την Δανέζικη Προεδρία να λάβει συγκεκριμένη στάση έναντι αυτού του φακέλου που είναι τόσο σημαντικό για του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Το Συμβούλιο. Εκπρόσωπο τη Προεδρία θέλει το λόγο, παρακαλώ. Για λίγο όμω περιορισμένο χρονό. Ευχαριστώ. Θα είμαι πραγματικά σύντομο η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε αίσιο πέρας σε αυτές τις συζητήσεις. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι θεμελιώδες επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα Σέγγεν θα πρέπει να συνεχίσει να ε, χαρακτηρίζεται από ισορροπία σε αυτό το τομέα και θα πρέπει να ενισχυθεί. Ελπίζουμε να επιτύχουμε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο για αυτή την πρόταση για τον κώδικα συνολών ώστε να λάβουμε εντολή ε, για την έναξη διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Καταγράψαμε τις θέσεις ε, των εκπροσώπων του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα και βεβαίως θα τις λάβουμε αυτές τις θέσεις υπόψη κατά τις εργασίες μας στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία βέβαια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Λίγα σύντομα σχόλια. Κοιτάξτε, είμαι ανοιχτή για να εξεύρουμε μία συμβαστική προσέγγιση, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά, να επιτύχουμε πρόοδο, προστατεύοντας όμως το σύστημα Σέγγεν. Εγώ θέλω να σας το πω και να σας Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλω το όνομά μου και την υπογραφή μου σε ένα αποτέλεσμα που θα σημαίνει υπονόμευση του Σέγγεν και α, μείωση των σημερινών προτύπων. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Ευχαριστώ κυρία Βέβερ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ψηφοφορίες. Τρεις ε, γνωμοδοτήσεις, συγγνώμη, τρεις εκθέσεις ε, θα πρέπει να περάσουν ψηφοφορία και μία ψήφος προσανατολισμού για την οδηγία για τις ε, συνθήκες υποδοχής των υπηκών των κρατών. Αρκετά μακροσκελής ο κατάλογος ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ να προετοιμάσετε τις ε, κάρτες σας. για να μπορέσετε να ψηφίσετε γρήγορα. Um, let's uh, start the vote. Ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και Νορβηγίας για την εφαρμογή σύμφωνων διατάξεων της Σύμβασης ε, του 2000 για την αμοιβαία αρρωγή σε ποινικέ υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο του 2001. Ο κύριος Μωράης θέλει το λόγο. Αν όχι, να περάσουμε άμεσα στην ψηφοφορία. Δεν υπευλήθη καμία τροπολογία. Άρα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος υπέρ. One vote. Okay, then we have to... Με συγχωρείτε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, όπως μου λέει η γραμματεία. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Αντζαλίλη, όχι, δεν έχω λάβει ακόμα την κάρτα μου. Θα προσθέσω το όνομά σας. Την κυρία Αντζελίλη. Την περιμένω, λέει κυρία Αντζελίλη, την κάρτα μου. Ούτε εγώ έχω την κάρτα μου, λέει κάποια άλλη συνάδελφος. Καταγράψτε δύο συναδέλφους. But we will, we might need uh, for the next Mrs. Lunacek. Κυρία Λουνατσέκ. Κυρία Λουνατσέκ. Μπορείτε να ζητήσετε από το βοηθό σα την κάρτα. Πέρασε ψηφοφορίας. Θα προσθέσουμε και μία ψήφο υπέρ. Άρα, 44 ψηφίσατε. 45 μάλλον ψηφίσατε. 45 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχέ. Συγχαρητήρια κύριε Μωράη. Next item. Το ερώτημα για την προφορική απάντηση τη Επιτροπής για το πράσινη Βίβλο για το δικαίωμα στην επανένωση οικογενειών των υπηκών των κρατών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Σαράντα πέντε υπέρ. Κανένας κατά δύο αποχές. Συγχαρητήρια. Εγκρίνεται λοιπόν. The third issue to be voted today. Το τρίτο που ψηφίζουμε σήμερα είναι η ψήφος προς προσανατολισμού. Okay, so please check it. Okay, uh, now the orientation vote on the. Ψήφος προσανατολισμού για τη σχέδιο έκθεσης που αφορά την οδηγή για τις συνθήκες εισόδου και διαμονής των επικών τρίτων κρατών στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής μετάθεσης. Εισηγητής ο κύριος Γιακολίνο. Τροπολογία 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτετα. 88. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι υιοθετείται λέει η πρόεδρος «91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Θέλω να το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay, I open the vote again. Closed. Λήξη ε, εντάξει. Δεκαέξι υπέρ, 33 κατά, καμία αποχή, οπότε απορρίπτεται 92. Υπέρ, κατά, αποχή, απορρίπτεται. 93, δεν θα ψηφιστεί σήμερα. Το 22 υιοθετείται χωρίς ψηφοφορία. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Πάμε στην το 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Α, έλεγχος για την 24. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 υπέρ, 28 κατά. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Employment 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 102 υπέρ. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Με αυτή τη συμβαστική καταπίπτουν άλλες τροπολογίες ε, στη συνέχεια του κειμένου. Πάμε στην τροπολογία 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Employment 31. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Ταυτόσιμη με τα 132. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε λοιπόν εκεί. Employment 32 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. Ταυτόσουμε με τα 133 και 134. Πάμε λοιπόν στην 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται σαφώς. Μετά 139 και εμπλέμε 34 επέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, αλλά θα ε, το ελέγξουμε. Ένα της ψηφοφορίας. Πέρας. 24 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο τελικά. Να πω μόνο ότι έχω τώρα την κάρτα μου, Πρόεδρε. Εντάξει. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Πέρα. 35 υπέρ, 15 κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σας ψηλά, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω. Τροπολογία 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Κύριε Αντζελίλη. Βάλτε το άλλο μηχάνημα. Εντάξει. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική υπέρ. Υπέρ. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 152 καταπίτη. Τροπολογία 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 καταπίπτει εξαιτία τη συμβαστική 6. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Employment 35 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 35 απασχόλησης. Τροπολογία 35 της Επιτροπής Απασχόλησης. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Και πάλι παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε νομίζω. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 167 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Έναρξη. 167. Πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 20 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 24 κατά. Υιοθετείτε, λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά είναι δύσκολο. Συμβαστική 10 υπέρ. Συγγνώμη, 170 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο νομίζω, άρα υιοθετείτε και πάλι. Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 170. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 25 υπέρ, 24 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. Εντάξει, 26 υπέρ. Α περάσουμε στην συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να πω, οπότε ας το ελέγξουμε. Έναρξη για την 177. Πέρα ψηφορία 27 υπέρ, 24 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. Έχουμε τέσσερι ταυτόσιμε ε, τροπολογίες. Επλώμε 36, 178, 179 και 180. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Υιοθετείτε. Η 181 καταπίπτει. 182 υπέρ κατά αποχές απο... απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Πάμε στην 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. 193 διορθώνει πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Περάς ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 24 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. Τον 94 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 και 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 202. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Πάμε στη 206 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι υιοθετείται. 215 υπέρ, κατά, το Υιοθετείτε. 216 υπέρ κατά ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 216. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.17. Θα ψηφίσουμε και το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας ή για το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε νομίζω. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίτεται. 18 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, για το 18. 24 υπέρ, 23 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. 2, 20 υπέρ. Κατά αποχές. Το ίδιο θα είναι νομίζω το αποτέλεσμα. Ας το ελέγξουμε 220. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 22 κατά. Υιοθετείτε λοιπόν. 19 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 20 υπέρ, κατά, Αποχές. Υιοθετείτε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τροπολογία 223. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στη 221. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας στη 224. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ 25 κατά. Υιοθετείτε. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω διοθετείτε. 2.26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. 2.26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι υιοθετείται. Ας ελέγξουμε για την 22. Εντάξει, υιοθετείται. 14. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 230. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε λοιπόν για τη 230. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Λήξη ψηφοφορία. 27 υπέρ, 21 κατά. Υιοθετείτε. «231 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για 37. Πάμε στη 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Περνάμε στη 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Και τώρα περνάμε μερικές σελίδες και φτάνουμε στη 280. Εντάξει. 280 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καταπίπτει η επόμενη και... 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προσχόληση 1 και τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προσχόληση 2 και 31 υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 3 και 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 και 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 επέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 πέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι οθετείτε, αλλά θα ελέγξουμε. Παρακαλώ ψηφίστε για τα 35. Πέρας ψηφοφορίας. 27 επέρ, 24 κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 καταπίπτει. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. τα 7 και τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για τη 43. Πέρας για τις 43 μιλούμε, 27 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. 44 και 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Της απασχόλησης 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά ας κάνουμε παλήθευση αρχίζει τροπολογία 1 πέρας 26 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται σε 9 και 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αυτή. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 12 όχι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 Επιτροπής Απασχολήσεως υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Εκπίπτει λοιπόν αυτή. Η 59, αυτή ψηφίζεται. 59 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60, 66, Α, πρέπει να ψηφίσουμε την 64 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση παρακαλώ, ακούγεται μια φωνή. Αρχίζει λοιπόν. 67 έτσι είναι. ...26 υπέρ 25 κατά. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εβδομήντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται αυτή. Τροπολογία 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά. Νομίζω ότι κρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αφήνουμε τη 16, 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά περνούμε στην 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχολήσεως 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση Πέρας. 38 υπέρ, 10 κατά. Δυστυχώς δεν είχατε σηκώσει τα χέρια σας. 84 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 απασχολήσεως υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 και 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το κείμενο ως ετροποποιήθη και αυτό θα το κάνουμε ονομαστικά, δηλαδή με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. «42 υπέρ, 5 κατά και 3 αποχές Συγχαρητήρια. Ακούστε παρακαλώ. Προχωρήσαμε ε, με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι προβλέπετο και ο διευθυντής της Frontex δεν έχει ακόμη φτάσει, άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. πριν από την ώρα που προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή 11 και 30. Well, 20 minutes before. I thought the vote would be much longer. Dear colleagues, uh, as, uh, as Mr. Lightning... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αφήχθη νωρίτερα ο κύριος Αντερμάν, ο κύριος Λάιτιν, συγγνώμη, και αν συμφωνείτε κι εσείς να συνεχίσουμε άμεσα τις εργασίες μας. Σημείο 26 της ημέρησης διάταξης. Έχουμε την παρουσίαση που θα μας κάνει ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της Frontex, ο κύριος Ιλκα Λάτινεν, για το πρόγραμμα εργασία ε, της Frontex. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κανονισμός ε, του Frontex τροποποιήθηκε πέρυσι, ο εισηγητής μας ήταν ο κύριος Μπουσουτήλ, και καλούμε τον κύριο Λάτινεν σήμερα να μας παρουσιάσει την Επιτροπή μας πώς πρακτικά θα τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις του κανονισμού και πώς αυτό θα τεκατοπιστεί στο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον Γκλάντιν και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη για α, συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και καλώς ήρθατε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να καλημερίσω τους αγαπητούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, είναι πάντοτε τιμή για μένα να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας. Πράγματι, θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2012. Δράτομαι όμως και της ευκαιρία, για να σας δώσω και μια απεικόνηση της παρούσας κατάστασης και τι νέα μας φέρνει η τροποποίηση του κανονισμού για τον οργανισμό μας. Να ξεκινήσω από την κατάσταση που της προηγούμενης χρονιάς, το 2011, χαρακτηρίστηκε από την Αραβική Άνοιξη. Αυτό ήταν το κυρίαρχο γεγονός. Σε ό,τι αφορά τις παράνομες διαλέψεις συνόρων προς την Ιταλία, είδαμε μία αύξηση 13 φορές περισσότερο σε σχέση με το 2010 για να σας δώσω μια εικόνα του όγκου. Κάτι άλλο σημαντικό είναι τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Αν δούμε τις τάσεις σε σχέση με το 2010, το 2011 παρατηρούμε μία μείωση πάνω από 30% σε αυτά τα σύνορα. Παρά τα αυτά, τα αριθμητικά στοιχεία παραμένουν σχετικά υψηλά. Κάτι άλλο που βλέπετε, στο στενό του Γιβραλτάρ, Είχαμε μία αύξηση προς την Ισπανία κατά 69% σε σχέση πάντοτε με το 2010. Οι δευτερεύουσες ροές που στήσαμε και πέρυσι αφορούσαν καταστάσεις ε, που είχαν οξυνθεί και να πόρνουν και Στη Ρουμανία είχαμε πενταπλάσια αύξηση των παράνομων τελέσεων σύνορων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και στην Ουγγαρία συν 50% η αύξηση. Έτσι για να σας δώσω μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Αν δούμε τώρα τα αριθμητικά στοιχεία, σύγκριση 2010 με 2011, βλέπουμε σαφώς ότι το 2011 είχαμε σχετικά αύξηση σχέση με το 10 ε, για τους λόγους που εξηγήσαμε. Είναι ενδιαφέρον επίσης να αναφέρουμε σε σχέση με 141.000 και συγκρίνουμε αυτό το στοιχείο με τις παρνόνιμες διαλέψεις στα συνοριακά σημεία διέλευσης που ήταν μόλις 300, 300 διαλέψεις, βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στην κατάσταση στα συνοριακά σημεία αδιαέλευσης και τα σημεία εισόδου. Κάτι άλλο που παρατηρήσαμε πέρυσι αφορά τις αρνήσεις εισόδου. Το 2011 η πλέον απαντόμενη ηθαγένεια ήταν αλβανή υπήκοη που τους αρνήθηκε η ενώ τις προηγούμενες χρονιές η πρώτη ε, υπηκότητα ήταν των Ουκρανών. Συγκρίνοντας λοιπόν αυτό, μιλάμε για συν 35% αύξηση ανάμεσα στο 10 και το 11 και ε, ενδιαφέρον ήταν ε, να παρατηρήσουμε ότι η κατανομή ανάμεσα στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα ήταν περίπου ισότιμη, 50-50. Στα χερσαία σύνορα είχαμε μία μείωση κατά 22%, ενώ στα θαλάσσια σύνορα η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην κατάσταση που αντιμετώπισε η Ιταλία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ο αριθμός των διευκολυντών. 21% λιγότεροι σε σχέση με το 10. Αυτό εν μέρη εξηγείται από τη μεγάλη πίεση που δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούσαμε. Οι βασικές εθνικότητες είναι περίπου ίδιοι. Αλγερινοί, που μπαίνουν πλέον στις πρώτες πέντε θέσεις, και Νιγύριοι. Μιλώντας για την Ιγυρία, να σας ενημερώσω με χαρά ότι στις 19 Ιανουαρίου η διευθέτηση ανάμεσα στις υπηρεσίες αλληλοδαπών της Νιγηρίας και τη Frontex υπογράψαμε μια σχετική συμφωνία. Η Αραβική Άνοιξη. Να διατέξω γρήγορα την κατάσταση, διότι είναι μια δυτή κατάσταση. Εστιάσουμε το θέμα στην Κεντρική Μεσόγειο συνολικά 65.000 ε, άτομα που αφορά την Ισίους κυρίως στην αρχή και άτομα που ε, έφυγαν από τη Λιβύη μετά την αρχή των εξεγέσεων. Τα στοιχεία στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι περίπου τα ίδια. Πάω τώρα στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Παραμένει δύσκολη κατάσταση και βλέπετε εκεί τη διακύμανση που είναι παρόμοια σε σχέση με το 2010. Αξίζει να σημειώσουμε ότι με τη βοήθεια των επιχειρήσεων Rabbit και την χερσαία επιχείρηση Ποσειδών, το ποσοστό ταυτοποίησης των προβλημάτων φτάνει το 90%. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μάλλον ότι εντοπίζονται σχεδόν όλες οι παρανομές διαλέψεις συνόρων. Έπειτα το ποσοστό του screening, δηλαδή οι ε, πρώτες συνεντεύξεις των παρανόμων μεταναστών ξεπερνά το 90%. Αναρωτάται λοιπόν κανεί γιατί τα αρνητικά στοιχεία είναι τόσο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο εντοπισμό και έχει γίνει η πρώτη συνέντευξη. Το πρόβλημα δεν αφορά το δυναμικό στον συνορικό έλεγχο, αλλά τι διαδικασίε πριν και μετά τα σύνορα. Αναφερόμαστε δηλαδή στην εργασία με την Τουρκία που θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Μιλούμε για το δυναμικό υποδοχής και κράτησης, καθώς με την αύξηση της εισρωής Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο ο αριθμός των παρανόμων αστών που αφήνονται από αυτά τα κέντρα. Και βεβαίω είναι κέντρα που αντιμετωπίζουν ε, πρόβλημα ε, για την καλή υποδοχή και κράτηση και αυτό αφορά επίσης και τον χρόνο της, ε, της κράτησης των ατόμων αυτών. Τώρα, για το χρόνο αντίδραση. Το 2011 ξεκινήσαμε μία επιχείρηση για ένα σχέδιο, το σχέδιο συγκυρίας της κατάστασης ήταν μια μεγάλη προσπάθεια που έπρεπε να κάνουμε, να λάβουμε υπόψη πολλά σενάρια και να λειτουργήσουμε έγκαιρα και προληπτικά. Ενισχύσαμε τις επιχειρήσεις στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα, στα focal points, όπως επίσης αυξήσαμε και το δυναμικό μας ε, στο επίπεδο των επιστροφών. Γι' αυτό η Δημοσιονομική Αρχή μας έδωσε 31,8 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, μπορούμε να δώσουμε μια σχετικά αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης και ένα μηχανισμό συνολικής παρακολούθησης της κατάστασης. Βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην εκτέλεση του προπολογισμού. Θα, θα σας πω λίγο λόγια για τον προλογισμό μετά σε ό,τι αφορά τον προλογισμό του 11, αλλά μία από τις συνέπειες ε, χρονική στιγμή που ήρθε η αύξηση του προπολογισμού ήταν ότι μας ανάγκασε να έχουμε σημαντικό υψηλό ε, κονδυλίων που μεταφέρθηκαν από το 11 στο 12. Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 36 εκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν. Ας πάμε τώρα στην εκτέλεση του προπολογισμού. Παρά ε, την προσθήκη του 31,8 εκατομμύρων ευρώ, μπορούμε να πω ότι ήταν υψηλό το ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού για το 10 είχαμε 69% το ποσοστό εκτέλεση του προπολογισμού, ενώ πέρυσι 66%. Να πω ότι ήδη στα τέλη του Σεπτέμβρη ήρθαν τα επιπρόσθετα 31 εκατομμύρια, οπότε πιστεύω τα πήγαμε αρκετά καλά. Το καλό νέο είναι πώς χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα που μεταφέρθηκαν από το 2010 στο προπολογισμό του 2011. Αυτά τα ποσά εκτελέστηκαν σε ένα ποστό 81%. Η συνολική λοιπόν εκτέλεση του προπολογισμού για τα πρώτα δύο χρόνια, ο προπολογισμός του 2009, εκτελέστηκε 182% και πέρυσι όταν ολοκληρώσαμε τη χρήση μεταφοράς, κατά 93% εκτελέστηκε ο προπολογισμός των χρημάτων του προπολογισμού του 10 χρησιμοποιήθηκαν και το 10 και το 11. Είναι σχετικά καλό αποτέλεσμα παρά το γεγονός για τους γνωστούς λόγους δεν καταφέραμε να τηρήσουμε απόλυτα τον ετήσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο προπολογισμό που τα χρήματα δαπανήθηκαν για τους σωστούς σκοπούς. Τώρα να περάσω στο 2012 που είναι και το αντικείμενο της παρουσίασής μου. Σε αυτόν τον χάρτη βλέπετε μία ε, καταγραφή τη ανάλυση κινδύνου που έχει κάνει η Frontex. Στο πιο σκοτεινό κομμάτι της διαφάνειας αφορά κυρίως τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Και βλέπετε από δυσμάς προς Ανατολάς, δηλαδή από το στενό του Βιγιαλτάρ, χωρί όμω να παραγνωρίζουμε τι Κανάριε νήσου, παρότι η εθνικά στοιχεία είναι πολύ, σχετικά μάλλον χαμηλά. Κυρίω εστιάζουμε στην κεντρική Μεσόγειο καθώς υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας και άρα υπάρχει, υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις εκεί. Βεβαίως και τα χερσαία σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας είναι σημαντικό θέμα για μας και τα σύνορα στα Βαλκάνια επίσης είναι σημαντικά για μας λόγω των δευτερογενών κινήσεων. Σε ό,τι αφορά τους αερολιμένες, σε αυτή την εικόνα στα πιο σκούρα κομμάτια, στις πιο σκούρες ε, χώρες, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας. Και τα βασικά αεροδρόμια που βλέπετε σε αυτό το χάρτη, στα οποία εστιάζουμε τις επιχειρήσεις μας, τα ενέργεια σύνορα, είναι ότι Βραζιλία, για παράδειγμα, είναι ε, χώρα που αντιμετωπίζει με τα προβλήματα. Η Αλγερία, η Νιγηρία, βλέπετε ότι έχουν πιο βαθύ χρώμα, Πακιστάν, Ινδία, ε, Κίνα και Ρωσία. Αυτές είναι οι χώρες στόχοι σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις για τα εναέρια σύνορα. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2012, περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ θα διοχετευτούν σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και πέρα από αυτά τα χρήματα, το υψηλότερο ποσοστό των χρημάτων που μεταφέρθηκαν από το 2011 στο 2012 θα διοχετευτούν σε αυτές τις δράσεις. Ελπίζω να βλέπετε τη διασύνδεση ανάμεσα στην προηγούμενη ε, διαφάνεια με τις περιοχές με το βαθύ χρώμα και σε αυτή τη διαφάνεια με τις κοινέ επιχειρήσεις. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα των κοινών ευρωπαϊκών ε, περιπολιών που συμπεριλαμβάνουν πολλές ε, θαλάσσιες επιχειρήσεις, ε, το έρασης και ε, στις νήσους, Μινέρβα στο ε, Γιβραλτάρ και ενίας στην περιοχή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Βεβαίως, ο Ποσειδώνα ε, στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα είναι πολύ σημαντική. Επίση, υπάρχει το project Attica για την αύξηση δυναμικού που προσπαθεί να στηρίξει την Ελλάδα ώστε να βελτιώσει τις ικανότητες που έχει ε, όσον αφορά τη διευθυντική των επιστροφών. Επίσης, κοινέ επιχειρήσεις Jupiter και ε, Neptune για τα χερσαία σύνορα μαζί με τι επιχειρήσει των focal points. Πρέπει να αναφέρω επίσης εδώ ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ε, που αναφέρουμε με κωδικές ονομασίες είναι επιχειρήσεις που περιέχουν μια σειρά φάσεων που θα πρέπει να εξαρθούν μέσα στη χρονιά βάσει της ανάλυσης κινδύνου που έχουμε κάνει. Πέρα από αυτό, προετοιμαζόμαστε να υλοποιήσουμε και εν μέρει ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση του επιχειρησιακού πακέτου ε, της ε, συγκυριακής κατάστασης και εδώ θέλω να πω ότι έχουμε 9 εκατομμύρια ευρώ αποθεματικό που μας έχει δώσει η Δημοσιονομική Αρχή ακριβώς για αυτό το σκοπό. Θα ζητήσουμε να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό στην περίπτωση που οι φυστάμενε επιχειρήσεις δεν επαρκούν. Στην περίπτωση που δεν θα μπορέσουμε να ιεραρχήσουμε εκ νέου τι προσπάθειές μας και αν λοιπόν όσα μπορούμε να κάνουμε δεν επαρκούν, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό. Κάτι άλλο που πρέπει να πω είναι η πρόσθετη πόρη για την εκπαίδευση και θα πω λίγα λόγια για αυτά. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, δαπανώνται για δραστηριότητες εκπαιδεύσεως. Εκτός από αυτές τις επιχειρήσεις, χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες, οι, αυτές που αναφέρονται στην επανεισδοχή είναι σημαντικές. Και εκεί έχουμε διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνουν 35 με 45 κοινέ επιχειρήσεις επιστροφής των ε, παρανόμων και σε διάφορους προορισμούς. Ελπίζω ότι αυτό πάλι εδώ συσχετίζεται με τη διαφάνεια όπου βλέπετε τις τρίτες χώρες που ε, αφορώνται εν προκειμένου. Και δύο λόγια τώρα για την επιχείρηση contingency plan, να σας δείξω δηλαδή την διάρθρωση αυτής της επιχείρησης. Βέβαια δεν είναι νέα, είναι επιχειρησιακές δραστηριότητες που ορισμένες από αυτές συνεχίζονται, άλλες ενισχύονται με τεχνικά μέσα ή με εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, ορισμένα από τα τμήματα αυτής της επιχειρήσεως contingency plan γίνεται, όπως για παράδειγμα η επέκταση της ε, επιχείρησης Ερμής ή επίσης η ενίσχυση του Ποσειδώνος και ούτω καθεξής. Τώρα, για την ε, ανάπτυξη δυναμικού, για τη δημιουργία ικανότητας, σαν capacity building. Γνωρίζετε ότι έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σχετική πρόταση και είναι προτεραιότητα του οργανισμού μας. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης που μας ε, μας απασχολεί πολύ και η δημιουργία pool ομάδων δηλαδή που προβλέπεται από το νέο τροποποιημένο κανονισμό με μεθοριακούς φρουρούς αλλά και τεχνικούς θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί και βέβαια για να ε, εξασφαλίζουμε και την τήρηση της υποχρέωσης αναφοράς. Ο τροποποιημένος κανονισμός περιλαμβάνει και πολλά σχετικά με την εκπαίδευση των ομάδων μεθοριακών φρουρών και εμείς ε, κάνουμε την εφαρμογή. Τώρα, δίνουμε και ιδιαίτερο βάρος σε αυτόματους ελέγχους των μεθορίων. Χορηγούμε επαγγελματική, ε, επαγγελματικές συμβουλές αλλά και πρακτική ενίσχυση για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων και, κυρίων, και κυρίως τα εισόδου-εξόδου με την τεχνολογική εξέλιξη των εφαρμογών που θα προχωρήσουν ε, για να δημιουργηθεί μια εικόνα ολόκληρης ευρωπαϊκής κατάστασης και το CPIP που είναι ε, η εικόνα που δίνεται πριν από τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση έχουμε τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η σταδιοδρομία των μεθοριακών φρουρών, η εκπαίδευση, τα προγράμματα εκπαίδευσής τους, ε, ένα είδος έρασμος και βέβαια μετά τα υψηλότερα επίπεδα σπουδών, με επίπεδο μάστερ κλπ. Εκεί δουλεύουμε σκληρά για να εναρμονίσουμε και να τυποποιήσουμε την ευρωπαϊκή εκπαίδευση μεθοριακών φρουρών. Το δεύτερο έχει σχέση με την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση. Εδώ τονίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε ένα πακέτο εκπαίδευσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνεργαζόμαστε με τους στρατηγικούς μας ε, εταίρους, με τον Υπατορμοστή ε, τον, ε, για τους πρόσφυγες και με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ και επίσης για τα θέματα πλαστών εγγράφων, σωματεμπορίας με τις αρχές του και λοιπά Αυτά όλα από το του δικού μας υλικού και χρησιμοποιούνται και από τους δικούς μας εκπαιδευτές. Ένα νέο στοιχείο που συζητείτε τώρα είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, ETS, European Training Scheme, για τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά επειδή έχουμε και πολύ στενές διασυνδέσεις με, την, με τις υπηρεσίες επιβολή του νόμου, αναπτύσσουμε το σύστημα αυτό ETS προς την κατεύθυνση αυτή. Και όταν έρχομαι στον προπολογισμό, τον φετινό, Μίλησα για το αποθεματικό των 9 εκατομμυρίων, για τους όρους για τον κεντρικό προϋπολογισμό. Για τρίτη χρονιά έχουμε μια πτωτική τάση του ε, προϋπολογισμού, όχι βέβαια τόσο δραματική, αλλά πάντως είναι ένας προϋπολογισμός που μειώνεται. Πέρσι ήταν εξαίρεση ή τα πρόσθετα εκείνα 31,8 εκατομμύρια ευρώ. Μίλησα και για τις μεταφορές από το 2011 για φέτος που ανέχονται σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση λοιπόν είναι επαρκής. Το μέγα πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η χρηματοδότηση. Το αποθεματικό είναι σημαντικό για να μπορούμε να είμαστε ε, σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και έχουμε βέβαια και ένα περιθώριο δημοσιονομικό ένα μέρος του επιχειρησιακού προϋπολογισμού της Frontex καταβάλλεται στις χώρες οι οποίες είναι χώρες υποδοχής των επιχειρήσεων. Μειώνουμε την τάση αυτή βέβαια, αλλά πάντως είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα μέσα στον οργανισμό. Η τάση είναι μείωση των χρημάτων που καταβάλλονται στις χώρες υποδοχής. Θα πρέπει να είναι οι εθνικοί προϋπολογισμοί και άλλοι μηχανισμοί και να χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτοί για τις συμμετέχουσες χώρες οι οποίες προσφέρουν εμπειρογνώμονες καθώς και τεχνικά μέσα. Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει βέβαια και πολλά νέα καθήκοντα που δεν θα τα αναφέρω αλλά υπενθυμίζω ότι όπως και φέτος το πρώτο εξάμεινο ο προϋπολογισμός της Frontex θα τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση της αρχής του προϋπολογισμού και μιλούμε για πρόσθετους ανθρώπινους πόρους για την κάλυψη θέσεων που απαιτεί ο νέος τροποποιημένος κανονισμός. Μιλούμε για περιορισμένο μάλλον αριθμό μελών, νέων μελών, μεταξύ 10 και 15 ε, προσώπων δηλαδή, εκεί, εκεί περίπου μιλούμε, για τόσα μιλούμε, και έρχομαι τώρα στον τροποποιημένο κανονισμό Frontex εμείς έχουμε δύο κατηγορίες εν προκειμένου. Η πρώτη κατηγορία είναι must και η άλλη είναι may. Ε, υποχρεωτικά και τα δυνητικά, ας πούμε, στοιχεία. Θα πρέπει να αρχίσουμε με αυτά που είναι υποχρεωτικά, μέτρα δηλαδή τα οποία έχουν σχέση με τις ομάδες μεθοριακών φρουρών, το Συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, εργαζόμαστε επ' αυτού, η διαδικασία κινείται προς μια κατεύθυνση όπου αμέσως μετά από το καλοκαίρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Μιλούμε για την σύνθεση τώρα, συζητούμε τη σύνθεση δηλαδή των αριθμό των συμμετεχόντων και ένα από τα ζητήματα εδώ είναι βέβαια να επιλεχθούν οι εκπρόσωποι του συνόλου των οργανώσεων ε, που ασχολούνται με τα θεμελίωτα δικαιώματα, μη κρατικέ οργανώσει κλπ. Ο διορισμός επίση ενό αξιωματούχου αρμοδίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι επίση ένα σημαντικό θέμα. Για την ώρα το οργανόγραμμα του 2012 δεν προβλέπει τέτοια θέση. Ωστόσο είναι κάτι που θα χρειαστούμε στο οργανόγραμμά μας για να εκπληρωθούν και τα όσα προβλέπει ο τροποποιημένος κανονισμός. Και βέβαια καλούμαστε να αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχετικά με τον εξοπλισμό και με τους αξιωματούχους οι οποίοι συμμετέχουν στα διάφορα πουλ ως προσκεκλημένοι να καθορίσουμε τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου αριθμού ε, μέσων τεχνικού εξοπλισμού για τις κοινέ επιχειρήσεις και Αυτά θα γίνουν όλα φέτος για το 2013 και μετά η ανάλυση του κινδύνου και μαζί με την ε, αξιολόγηση των ικανοτήτων των χωρών μελών. Αυτά θα γίνονται επίση σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς φέτος συζητούμε τα κριτήρια, τους τρόπους αξιολόγησης των ε, ικανοτήτων των χωρών μελών. Η αγορά και η μίσθωση εξοπλισμού. Κάνουμε τα πρώτα βήματα για να δούμε κατά πόσον αυτό θα είναι απαραίτητο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ένα από τα κύρια σημεία του τροποποιημένου κανονισμού, εδώ εμείς εργαζόμαστε σκληρά για να φτιάξουμε την βασική υποδομή που θα επιτρέψει την διαφύλαξη της ακαιρεότητας των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης συζητούμε και τους τρόπους και όρους της ανταλλαγής και αυτά θα υλοποιηθούν το 2013. Επίσης η πρόσληψη ε, second guest officers που είναι επίσης πολύ σημαντική και το ίδιο είναι και οι αποστολές τεχνικής υποστήριξης σε τρίτες χώρες. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι όροι εν προκειμένου ποιος θα μπορεί να είναι ο όγκος αυτών των, επιχειρή... των ε, αποστολών και πώς θα εντάξουμε τι αποστολέ αυτές στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση, καθώς επίση και οι αξιωματικοί σύνδεσμοι και η σχετική πρόσληψη, η πρόσληψή τους δηλαδή, και σε τρίτες χώρες. Αυτά όλα σημαίνουν βέβαια ότι γνωρίζουμε βέβαια την δημοσιονομική κατάσταση, γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτική μηδενικής Αύξηση Έχουμε τον νέο τροποποιημένο κανονισμό και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και αναθεωρούμε μάλιστα τη στρατηγική του οργανισμού μας. Βλέπετε εδώ αριστερά τις αξίες του επαγγελματισμού και της ανθρωπιάς που εξακολουθούν να υπάρχουν και που βασίζονται στο ανοιχτό πνεύμα και στην συνεργασία η νέα μας στρατηγική θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην προστιθέμενη αξία. Ό,τι και να κάνουμε δηλαδή επιθυμούμε να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Ρίχνοντας ιδιαίτερο φως στις ικανότητες των χωρών μελών, διότι αυτές φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο των συνόρων. Έχουμε εντοπίσει πέντε ή έξι, έξι καλύτερα, κύριους στόχους στη νέα στρατηγική αφενός για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ε, χωρών μελών, δεύτερο η ορθή αντίληψη των ε, καταστάσεων, ενίσχυση της ανταπόκρισης, ανταπόκριση σε επίγουσες καταστάσεις και σχετικές επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένα θέματα οργανωτικά ή προσωπικού. Εδώ έρχομαι στο τέλος της ε, παρουσιάσεώς μου για το πρόγραμμα εργασιών και ευχαριστώ θα ακούσω τα σχόλια ε, που έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα. Συνάδελφοι, έχετε το, το λόγο τώρα, κύριε Μπουζόκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά, να ευχαριστήσω τον κύριο Λάτινεν για την παρουσίασή του Του εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ε, φετινή χρονιά που θα είναι πολύ σημαντική για τον Frontex, όχι μόνο επειδή ε, έχει τον προπολογισμό που ήθελε, αλλά και επειδή θα πρέπει να εφαρμόσει τον νέο κανονισμό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά τα δυνητικά στοιχεία που αναφέρετε θα γίνουν υποχρεωτικά για το 2012 και όχι το 2013. Εμείς ε, θα επιβλέπουμε την, και θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τη δράση ε, του Frontex και θα παρεμβαίνουμε όπου θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Να πω κάτι για τον προπολογισμό όμως. Ή, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα στήριζε τις ανάγκες ε, του οργανισμού σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και αν θυμάμαι καλά, ο αρχικός προπολογισμό ανερχόταν σε 20 εκατομμύρια, αν όχι λιγότερο. Και τώρα έχετε περίπου έχετε προπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ε, οπότε έχει επιληθεί το ζήτημα του προπολογισμού για σας. Μόλις χθε όμως, κύριε Λάιτινεν, αυτή η Επιτροπή συζήτησε την, και εξέτασε τη γνωμοδότηση για την απαλλαγή προπολογισμού για το 2010 ε, μεταξύ άλλων και για το δικό σας οργανισμό. Και τουλάχιστον για το δεύτερο ε, έτος δεύτερο συνεχόμενο έτος, ίσως και παραπάνω, παρατηρήσαμε την, ε, το μεγάλο αριθμό των μεταφορών carryovers. Είπατε σήμερα ότι το ίδιο θα ισχύσει και για το 2011. Όταν θα συζητήσουμε δηλαδή ε, την απαλλαγή και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα χαρεί καθόλου. Δεν ε, θα συμφωνήσει να δώσει απαλλαγή με μια τέτοια συνεχιζόμενη κατάσταση σημαντικής μεταφοράς ε, ποσών από τη μια χρονιά στην επόμενη. Ε, σας καλώ λοιπόν να επιλύσετε αυτή την κατάσταση μια για πάντα. Βεβαίως και κατανοούμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζετε, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιχειρησιακές με τα επιχειρησιακά καθήκοντα του οργανισμού που δεν είναι πάντα κάτι προγραμματισμένο. Κάποιες φορές ε, πρέπει να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που ανακύπτουν εκείνη τη στιγμή. Όμως φέτος η απαλλαγή θα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας αν συνεχίσουν αυτές οι υπερβολικές μεταφορές. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω αφορά Ε, της, ε, την διέλευση των συνόρων στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για μας παρά την ανάπτυξη των ομάδων Rabbits αυτής της αποστολής το 2010 και μετά με την ε, επιχείρηση Ποσειδώνας. Τα στατιστικά αρχικά έπεσαν και μετά ξανανέβηκαν και αν κατάλαβα καλά τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερα σε σχέση με πριν από την ανάπτυξη των Rabbits. Αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Θα ήθελα να μου δώσετε περαιτέρω πληροφορίες. Ποια είναι η δική σας πρόθεση. Η αντίδραση ήταν ότι αρχικά όλοι πίστευαν ότι τα σύνορα είναι κλειστά επειδή ήταν εκεί ο Frontex. Μετά όμως είδαμε ότι τα σύνορα δεν είναι κλειστά, ακόμα και αν είναι εκεί ο Frontex. Και αυτό και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε λίγο πιο αναλυτικά. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έφυγε, έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο, αλλά και αυτός θέλει να σας ε, θέσει ένα ερώτημα για αυτό το ζήτημα, γιατί ε, τον απασχολεί ιδιαίτερα. Μερικά ακόμα ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Πρώτα απ' όλα, το Συμβουλευτικό Φόρουμ είπατε ότι έχετε δυσκολίες στην ταυτοποίηση των οργανισμών που θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί ε, αυτά τα γνωμοδοτικά φόρα ε, έχουν συσταθεί από, άλλες, από άλλους οργανώσεις. μόλις τον περασμένο μήνα η άσο που είναι πολύ πιο νέα ηλικιακά εντό εισαγωγικών ε, σε σχέση με εσά, έκανε ήδη την πρώτη συνεδρίαση νομοδοτικού φόρουμ. Αν δείτε λοιπόν άλλου οργανισμού, θα δείτε ποιε διακεκριμένε οργανώσει ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, πέρα από τι προφανεί, ε, θα πρέπει να συμμετάσχουν. Τώρα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το αντίστοιχο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται στο γενικότερο πλάνο σας. Όμως, τι σας ε, εμποδίζει να το τροποποιήσετε και να προσλάβετε έναν τέτοιο υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ακόμα και να αναθέσετε σε κάποιο μέλος του προσωπικού σας αυτά τα καθήκοντα. Και αυτό μάλιστα το σημαντικό δυνατό. Η Επιτροπή μας λοιπόν πραγματικά θα ήθελε να λάβει αυτό το καθησυχαστικό μήνυμα ότι θα ε, διοριστεί κάποιος ε, τέτοιος υπεύθυνος. Τώρα για την συνεργασία με τρίτες χώρες. Αναφέρατε μία συμφωνία που υπεγράφει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με την Ιγυρία. Θα ήθελα να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες όμως ε, σε ό,τι αφορά άλλες χώρες. Για παράδειγμα, υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία με την Τινησία, την Αίγυπτο και, ή βεβαίω και με τη Λιβύη, που τώρα έχει ε, ε κάποιου είδους κυβέρνηση, παρόλο που ε, παραμένουν ρευστά τα πράγματα. Και βεβαίως ε, συνεργασία, η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο πρόγραμμά σας. Για τις ε, επιχειρήσεις επανεισδοχής μπορείτε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες. Εξετάζοντα το σχέδιό σας, ε, λέγατε ότι θέλετε να έχετε περίπου 30 τέτοιε αποστολές. Τουλάχιστον αυτές έχετε προγραμματίσει στον προπολογισμό. Δώστε μας ε, κάποιες πληροφορίες ακόμα. Πώς ακριβώ προτίθεστε να το κάνετε αυτό, γιατί τώρα έχετε το δικαίωμα πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα. Θα θέλαμε λοιπόν ο οργανισμός ε, μέσα στο 2012 να λάβει έναν ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή των ε, λάθρων μεταναστών που διαμένουν παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, για τις ε, ευρωπαϊκές ε, ομάδες μεθοριακής φύλαξης κάνει κάτι ο οργανισμός για τον σχεδιασμό σε αυτόν το τομέα. ουσιαστικά θα πρόκειται για άτομα που ήδη βρίσκονταν σε αυτή την ομάδα ή θα, θα κάνετε νέες προσπάθειες για να ενισχύσετε ε, την ήδη φυστάμενη ομάδα. Συγγνώμη αν σας φόρτωσα με πολλά ερωτήματα. Μάλιστα ε, άφησα και μερικά απ' έξω. Ελπίζω να έχετε μερικές απαντήσεις για μένα. Ευχαριστώ. Okay. Ε. Εντάξει, θέλετε να απαντήσετε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν γιατί ήταν πολλά τα ερωτήματα. Υπάρχουν τρεις ακόμα παρεμβάσεις. Ναι, αλλά είναι ήδη αυτά τα ερωτήματα. Συνήθως ακούμε όλες τις παρεμβάσεις και μετά ακούμε τις απαντήσεις σας, αν συμφωνείτε. Κυρία Ρομέρο Λόπες. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή του Frontex, ο οποίος μας έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αν μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς αυτή την παρουσίαση, θα ήταν πραγματικά ευχάριστο. Ναι, εντάξει τώρα, ακούτε τη διερμηνία. Παραλαμβάνει ο Μιλήτρια, ευχαριστούμε πολύ τις πληροφορίες, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο να λάβουμε και εμείς αυτή την παρουσίαση με τα δεδομένα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε αντίστοιχε παρουσιάσει ε, είχατε έρθει με κάποια έκθεση. Τώρα κάνετε μια πολύ πιο άμεση παρουσίαση. Θα ήταν σκόπιμο να την έχουμε. Παρόμοια ερώτηση με αυτή τη δέσμη των ερωτήσεων του κ. Μπουσουτήλ. Το σχέδιο με την Ιγυρία που μας ανακοινώσατε. Ο οργανισμός έχει την εξουσία να επιλέξει με ποιες χώρες προβλέπει να κάνει μια συμφωνία ή ένα σχέδιο. Και γιατί επιλέξατε την Νιγηρία. Ποιες ήταν οι δυσκολίες να κάνετε κάτι αντίστοιχο με τη Σομαλία, για παράδειγμα. Είναι η Σομαλία μία από τις χώρες που μας δίνει τους μεγαλύτερους αριθμούς το άσυλο. Το Αφγανιστάν επίσης. Η Τινησία, Λιβύη. Επίτασε τι συνίσταται αυτό το σχέδιο με την Ιγυρία. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια περισσότερα σχετικά με τις αρμοδιότητες εξουσίες που έχει ο οργανισμός για να ξεκινήσει αυτόνομα ως οργανισμός αυτή τη συνεργασία. Αυτόνομα λοιπόν πώς μπορείτε να ξεκινήσει συνεργασία με αυτές τις χώρες. Βεβαίως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και θα ήθελα να εμβαθύνετε σε αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Αφορά κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία που μας δώσατε σχετικά με τους παράνομους μετανάστες. και την κράτησή τους στα σύνορα. Αν κατάλαβα καλά, είναι πολύ ψηλό το... ο αριθμός τους. Μόλις 20.000 ήταν αυτοί που κατάφεραν τελικά να ξεγελάσουν τις αρχές και να μην τυχούν κράτηση. Είναι πολύ χαμηλός λοιπόν ο αριθμός αυτός που ξέφυγαν αν θέλετε. Μπορείτε να μου το δεικνύσετε. Αυτόν τον αριθμό των ε, μεταναστών που κατάφεραν να ξεφύγουν, να ξεγλιστρήσουν από το σύστημα. Είναι αριθμητικά στοιχεία που αφορούν μόνο τα εναέρια σύνορα, τα χερσαία, τα θαλάσσια, συνολικά. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Έπειτα, ένα άλλο αριθμητικό στοιχείο που αφορά του ετούντε άσυλο, 234.000 λέει ο Μιλήτρια είπατε. Πρώτα απ' όλα, πώ καταλήξατε σε αυτό το στοιχείο, γιατί χθε ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο, τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του Ασύλου στη Μάλτα και μας είπε ότι δεν έχει την ευχέρεια το γραφείο να λάβει τις κράτη-μέλη. Εμείς ρωτήσαμε πώς είναι τούτε άσυλο στα 27 κράτη-μέλη και μας είπε ότι δεν έχετε τέτοια στοιχεία και ότι το ε, Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου παίρνει πληροφορίες από ε, τις μη κυβερνικές οργανώσεις. Και ρωτώ, εσείς από πού αποσπατά τις πληροφορίες, πώς κάνετε αυτά τα συστατικά στοιχεία και συνέπεια αυτές τις ερώτηση, Αυτοί του άσυλο πού βρίσκονται. 234.000 ετούντες άσυλο Κάπου πρέπει να βρίσκονται. Είναι στα κέντρα κράτησης. Στα αριθμητικά στοιχεία που μας δώσατε, δεν μας εξηγήσατε κατά πόσον έλαβαν το καθεστώς του πρόσφυγα ή όχι. Αν όχι, ποιο είναι το ποσοστό εξ αυτών που παραμένει στα σύνορα περιμένοντας μία απόφαση στην αίτησή τους και σε τι είδους κέντρα βρίσκονται, σε ποιες χώρες. Πού είναι η μεγαλύτερη πίεση στις αιτήσει ασύλου. Και τέλος, τελευταία ερώτηση σχετική με αυτή που μόλις έκανα. Όταν κάνετε μια περιπολία με σκοπό να προβείτε σε σύλληψη στα θαλάσσια, χερσαία, αλλά ακόμα και στα νερία σύνορα, πώς διακρίνεται έναν ετούντα άσυλο από έναν παρόν μετανάστη. Ευχαριστούμε. Κυρία Κέλλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ με πολλά από τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα για τον ε, υπεύθυνο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα μπορούμε και από μόνο εδώ στα γρήγορα να σας πούμε ε, αρκετές τέτοιες οργανώσεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού έγινε το πρόβλημα. Αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για τον Human Rights Officer, αυτή η Επιτροπή εξέτασε τις, ε, ε, τις δημοσιονομικές διατάξεις και είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτά τα 80 εκατομμύρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή του νέου κανονισμού μεταξύ άλλων και για την πρόσληψη ενό ε, τέτοιου αξιωματικού υπευθύνου. Πρέπει να μου εξηγήσετε λοιπόν το ποιο είναι το πρόβλημα. Για τον νέο κανονισμό επίση ε, συμπεριλαμβάνει την ε, διάταξη ότι θα πρέπει ο Frontex να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις παράβασης και μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό συμβαίνει συστηματικά. Πολλοί μετανάστες ε, κρατούνται σε μη βιώσιμες ε, συνθήκες. Το γνωρίζετε αυτό. Κατά γνώμη, δεν, κατά γνώμη μου δεν έχετε κάνει κάποια... δεν έχετε φύγει από αυτή την αποστολή ακόμα. Το εξετάζετε το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε και σε τι θα ποια θα είναι η απόφασή σας περί αυτού. Μετά, για την μεταφορά ε, των κονδυλίων και αυτό δεν μου αρέσει γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μην ξανασυμβεί. Και τώρα βλέπουμε ότι ξανασυμβαίνει. Είπατε ότι 36 εκατομμύρια θα μεταφερθούν πάνω κάτω ή 31 και περίπου το ίδιο ποσό ήταν τα, τα επιπλέον κονδύλια που σας ε, δόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι πάνω κάτω λοιπόν το ίδιο, το, το, το ίδιο ποσό. Νομίζετε ότι αυτά τα επιπρόσθετα χρήματα δόθηκαν πολύ αργά. Τι ακριβώς συνέβη. Πώς χρησιμοποιήσατε αυτά τα επιπλέον κονδύλια. Γιατί υπάρχει έλλειψη ικανότητας απορρόφησης. Κανονικά θα πρέπει να είστε σε θέση να το απορροφήσετε κατευθείαν. Μετά, μας δείξατε τις χώρες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ζώνες ε, κρίσιμες χώρες για προέλευσης ε, μεταναστών, γυρία κτλ. Και επίσης αναφερθήκατε και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορείτε να εξηγήσετε και αυτό. Μετά για το αποθεματικό 9 εκατομμύρια είπατε ότι είναι. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του αποθεματικού. Έχω μερικές ακόμα, αλλά όχι πολλές. το EDPS ε, έκανε μια σύσταση στον Frontex για τα δικαιώματα ε, ε, των μεταναστών σε περιπτώσεις επανεισδοχής και δεν εφαρμόστηκε τουλάχιστον έως πριν με μερικές εβδομάδες. Θα μας ενημερώσετε για το αν έχετε εφαρμοστεί και αν όχι πότε θα το κάνετε και γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα. Αυτά. Το τελευταίο μου ερώτημα προς την Επιτροπή θα θέλω να το απευθύνω, γιατί έχει αναλάβει νέε ε, αρμοδιότητες. Δεν ξέρω ποιο είναι εδώ από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την, εποπτεία, την παρακολούθηση, είπαμε ότι θα, η Επιτροπή θα φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα ε, στις επιχειρήσεις επανεισδοχής. Θα μας ε, ενημερώσετε για το τι συμβαίνει εκεί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Κορτσέτα. Eh, ε, πριν ξεκινήσει το τέλος του Καντάφη, ο Frontex είχε δείξει μεγάλη ενεργητικότητα στη σύναψη μια συμφωνίας με τη Λιβύη για τον έλεγχο της μετανάστευση. Βεβαίω, αφού η Ιταλία δεν είχε κινηθεί, γιατί να μην το κάνει η Ευρώπη, το κατανοώ. Βεβαίω μετά είχαμε τις παγκόσμιες πολιτικές εξέλιξεις που αφορούν και πρόσωπα και η κακή τελικά μοίρα του δικτάτορα οδήγησαν σε αυτούς που υποστήριζαν της, ε, τη συνεργασία με τέτοιες εγκληματικές προσωπικότητες με τελικά να παίρνουν τις αποστάσεις τους. Ξέρετε υπάρχει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Τομάς του Λεμπετούσα, ο Κατόπαρδος, που τελικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τελικά κάνουμε πάρα πολλά, καλάσουμε πάρα πολλά για να μην αλλάξουμε τίποτα. Πώς γίνεται λοιπόν, καταλήγουμε να προσφέρουμε την ίδια συμφωνία στην Λιβύη την μεταναστατική με την ίδια συμφωνία που είχαμε προσφέρει στον Καντάφη. Απορώ δηλαδή από άποψη κράτους δικαίου πώς κάνουμε την ίδια πρόταση. Ιδίως μετά τις καταγγελίες που έγιναν για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την εποχή του κατάφη έναντι των μεταναστών, άτομα που υπέστησαν βασανιστήρια, γυναίκες που ε, έπεσαν θύματα βιασμού στα κέντρα υποδοχής στη Λιβύη, όπως και άτομα που συνελήφθησαν στην ε, ε, έρημο προσπαθώντας να ξεφύγουν από κέντρα κράτηση στη Λιβύη. Να πω κάτι άλλο τώρα. Η Μεσόγειος έχει καταντήσει μία, ένα τεράστιο νεκροταφείο Ήμουν ε, δήμαρχος στην πόλη μου, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη, και σε ένα ναυάγιο είδα τα πτώματα 11 ανθρώπων, παιδιά 15, 16, 17, 20 χρονών, που πέθαναν ε, μέσα σε αυτά τα σαφρά πλοία που τους επιβιώσατε, τι παρατηρήσαμε ότι λαμβάνοντα υπόψη και ποια είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω λαμβάνοντα υπόψη και την Ιταλική νομοθεσία και πώ νοεί ω λαθρέου όλου αυτού τους ανθρώπου χωρί να έχει ταυτοποιηθεί η ταυτότητά του. Πολλά σκάφη αρνούνται να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και να τους αφήσουν να ανέβουν στο πλοίο. Άρα καταλήγουν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Frontex έχει εντάξει στο πρόγραμμά του μια ανθρωπιστική αποστολή. Αυτό πιστεύω ότι θα απέντε τα εύσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επέτρεπε με τον τρόπο να απομονώσουμε και κάποιες αυταρχικές φωνές που ακούγονται στην Ευρώπη πριν απορρίψουμε δεν πρέπει να διαπιστώνουμε κατά πόσον υπάρχουν πραγματικοί έτοντες άσυλο. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο α, των Ηνωμένων Εθνών, κάτι τέτοιο προβλέπεται. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται. Θα ήθελα ειλικρινά να καταλάβω καλύτερα ποιες είναι οι πολιτικές γραμμές ε, που προτίθεται να ακολουθήσει η Frontex. Ευχαριστώ κύριε Κροτσέτα. Να δώσω τότε το λόγο στον ε, κύριο Λάτινεν και πάλι να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω όχι απλά να προσπαθήσω, αλλά και να καταφέρω να απαντήσω. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για τα ερωτήματα. Ε, Πράγματι, δεν ε, έδωσα πάρα πολλέ λεπτομέρειε στην παρουσίασή μου. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τι μεταφορέ των κονδυλίων από το ένα έτο στο άλλο. Η φύση των δραστηριοτήτων που διεξάγει η Frontex μας αναγκάζει να έχουμε πάντοτε τέτοιες μεταφορές και μάλιστα μιλούμε για υψηλά ποσά που μεταφέρονται. Βεβαίω, υπάρχει μια θετική εξέλιξη και θέλω να σα εξηγήσω το γιατί οι επιχειρήσει βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου. Κάποιες επιχειρήσει ξεκινούν αρκετά αργά μέσα στο έτος. Άρα τι σημαίνει. Όταν ολοκληρωθεί η επιχειρησιακή φάση, μπορούν να τύχουν επεξεργασία τα τιμολόγια. Και ο χρόνος επεξεργασίας πολλές φορές ξεπερνά το ίδιο μυρολογιακό έτος. Άρα είναι καλύτερο να βλέπουμε συνολικά το χρόνο ε, υλοποίησης, άρα αναδιατία. Βεβαίω προτεραιότητα είναι να χρησιμοποιούμε και να εκτελούμε τον προπολογισμό ετησίω. Μην με παρερμηνεύετε. Ο στόχος είναι να εκτελούμε τον προπολογισμό μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Αν όμως ε, έτος 1 συν 10 και μετα... δούμε συνολικά τα ποσά που μεταφέρονται και δούμε αν αυτά τα χρήματα που μεταφέρονται χρησιμοποιούνται την επόμενη χρονιά, εκεί είναι η ουσία. Γι' αυτό σας έδωσα τα στοιχεία του 2010, του προβλογισμού του 10, όπου είχαμε ένα σχετικά υψηλό αριθμό μεταφορών και μετά το 11 επιτύχαμε 93% εκτέλεση του προπολογισμού. Και δηλώνω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Άρα καταφέρεμε να χρησιμοποιήσουμε ορθά και για τον καλό σκοπό τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Όχι μεν απόλυτα στο έτος, στο οικονομικό έτος το οποίο προβλεπόταν, αλλά στην επόμενη χρονιά. Τώρα, ε, για φέτος που έχουμε τα 36 εκατομμύρια που μεταφέρθηκαν στην επόμενη χρονιά, είναι ότι όταν ξεκινά μια επιχείρηση, δεν μπορεί να ξεκινήσει η επιχείρηση πριν ε, καταγραφούν αυτά τα χρήματα στο προπολογισμό. Οπότε αυτά τα επιπλέον 36 εκατομμύρια δεν υπήρχαν στο προπολογισμό του Frontex πριν τις αρχές Οκτωβρίου. Άρα δεν είμαστε σε θέση να προβούμε σε ανάληψη της υποχρέωσης. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε την ανάληψη υποχρέωσης, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα προπολογισμού και άρα δεν δεσμεύονται και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στην επιχείρηση. Πρέπει να περιμένουμε από τη χρονική στιγμή όπου λαμβάνεται η απόφαση για τον προπολογισμό, εγγράφεται το ποσό στον προπολογισμό, οπότε τότε μπορεί να αναλυφθεί η υποχρέωση και τότε μπαίνουν και τα κράτη-μέλη στη διαδικασία τη συμμετοχή. Και παρατηρούμε ότι η διαδικασία τροποποίηση του προπολογισμού και αυτή είναι χρονοβόρα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, για το 2012 και ελπίζω και εφ' εξής, υπάρχει αυτό το αποθεματικό, θα υπάρχει το αποθεματικό και θα είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιούνται τα χρήματα του αποθεματικού όταν υπάρχει ανάγκη για γρήγορη χρήση κονδύλιων. Άρα το θέμα δεν είναι κατά πόσον είναι ε, ορθή ε, η δημοσιονομική διαχείριση, κατά πόσον τα χρήματα χρησιμοποιούνται ακριβώς για το σκοπό για το οποίο έχουν δοθεί. Δεύτερο, προς τον κύριο Μπουσοτήλ για τα χερσαία σύνορα της Τουρκίας. Ανέφερα δύο αριθμητικά στοιχεία που ξεπερνούν το 90%. Το ποσοστό εντοπισμού και ποσοστό πρώτων συνεντεύξεων. Και έπειτα, λέμε, είπατε τι άλλο μπορούν να κάνουμε θεωριακοί φρουρή στόχος είναι να αποφευχθούν οι λαθρές διαλέψεις. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, αυτό είναι ερώτημα. Αν ο παρανός μετανάστης θέλει να διέλθει των σύνορων, πολύ απλά διέρχεται τα σύνορα. Εντοπίζεται, συλλαμβάνεται και μετά ξεκινά μια διαδικασία. Είτε υπάρχει διαδικασία ασύλου, άρα αρμόδιες είναι αρχές ασύλου, αν όχι, ξεκινά μία διαδικασία που έχει ως τελικό σκοπό την επιστροφή. Γι' αυτό έχουμε δύο διαδικασίες. Δεν είναι θέμα ικανότητας ε, ελέγχου των σύνορων, είναι κατά πόσο λειτουργεί όλο το σύστημα πριν φτάσουμε στα σύνορα. Γι' αυτό μίλησε για τη συνεργασία με την Τουρκία. Η διακύμανση που είδατε στο διάγραμμα είναι πιο πολύ εποχικού χαρακτήρα. Βλέπετε ποια είναι η στάθμη των υδάτων στον ποταμό ε, του Εύρου, η θερμοκρασία της εποχής κτλ. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις. Αν ε, έλεγα ένα πράγμα το οποίο μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση είναι θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δυναμικό για τον οντοπισμό και την, υποδοχή, και την ε, σύλληψη. Βεβαίω υπάρχει ανθρωπιστική πτυχή και όλοι την γνωρίζουμε. Αλλά αν είχαμε μεγαλύτερο δυναμικό εντοπισμού και σύλληψη, τότε θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα. Και για τη διαδικασία και για τη διαδικασία επιστροφή. Υπάρχουν με, παρόν μετανάστες που ενώ κανονικά πρέπει να τύχουν επιστροφή, τελικά α, α, αφήνονται από την κράτηση γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο δυναμικό. Πάντως εντοπίζουμε και κάνουμε την πρώτη συνέντευξη σε πάτο το 90% των παρανόμων. Σε ό,τι αφορά το συμβουλευτικό αυτό φόρουμ, ίσως να τα είπα τα πράγματα κάπως απεσιόδοξα. Η διαδικασία παρά τα αυτά πηγαίνει αρκετά καλά. Είναι ένα μάλλον θετικό πρόβλημα το που μας απασχολεί, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επί του θέματος. Θα πρέπει να βασιστούμε στο χρονοδιάγραμμα και όπως προβλέπει ο κανονισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για αυτό. Έχουμε πέντε συνεδριάσεις ετησίως και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε ποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται τι. Η επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 8 και 9 Φεβρουαρίου, οπότε θα συζητήσουμε το τεχνικό χρονοδιάγραμμα, αλλά και την σύνθεση του φόρουμ αυτού. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τον Οργανισμό Θεμελιών Δικαιωμάτων επί του θέματος και φυσικά έχουμε πολύ μεγάλη υποστήριξη και από εκείνη την πλευρά. Τώρα, ο υπάλληλο, ο υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε ε, ένα τέτοιο άτομο αν δεν προβλέπεται τέτοια θέση. Α, αν δεν έχει τροποποιηθεί επίσης ο προϋπολογισμός για να υπάρξει ειδική γραμμή για την ε, μια τέτοια θέση, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη θέση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δικασία για το διαγωνισμό, αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί η θέση. Πρέπει λοιπόν βάσει του κανονισμού πρώτα απ' όλα να τροποποιηθεί η σχετική γραμμή του προπολογισμού και εκεί είναι το πρόβλημα. Όμως υπάρχουν όλες οι προετοιμασίες, ε, υπάρχει το, το προφίλ της θέσης, έχει ε, προκηρυχθεί ε, η θέση Τώρα, για τις επιχειρήσεις επιστροφών. 35 με 45 επιχειρήσεις ετησίω. Δεν μπορώ να δώσω πολύ συγκεκριμένο στοιχείο γιατί είναι τέτοια η φύση ε, των επιστροφών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι να υπάρξει αποδοχή της επανεισδοχής στη χώρα επιστροφής και πολύ συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης των διπλωματικών οδών με αυτές τις τρεις χώρες. Εμείς δεν έχουμε αυτό το δυναμικό. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διπλωματικές οδούς και Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτέ τι κοινέ επιχείρησεις στα κράτη-μέλη. Εκεί τα κράτη-μέλη μπορούν να βοηθήσουν με τις διπλωματικές τους επαφέ και να επιτύχουμε καλύτερα τι επιστροφέ. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ε, και επιμελητία, αλλά πρέπει να διευθετούνται οι επιστροφές με τέτοιο τρόπο ώστε η χώρα υποδοχής να δεχτεί πρώτα απ' όλα την προσγείωση της πτήσης και να δεχτεί πρακτικά ε, τους, ε, τα άτομα αυτά. Τρίτε χώρες. Την Ισία και Λιβύη. Είχαμε επαφές και με τις δύο χώρες στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορούμε εμείς ως Frontex να προσεγγίσουμε αυτές τις χώρες. Δεν θα υπάρξει απάντηση από πλευρά τους. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές αποστολές. Από ό,τι γνωρίζω δύο αποστολές ε, έγιναν στην Τινησία, μία στην Λιβύη τουλάχιστον και άρα θα μέσω αυτών. Τουρκία. Προς το παρόν κανένα συνταρακτικό νέο. Αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στην πλευρά της Τουρκίας με τους διαπραγματευτές από τουρκικής πλευράς καταφέραμε να συμφωνήσουμε μία εκδοχή της διευθέτησης εργασίας. Τώρα υπάρχουν ιστορικές διαβουλεύσεις στην Τουρκία που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Και αυτό βεβαίως γίνεται ε, για κάθε εκδοχή όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο το ζήτημα. Δεν ε, αφορά μόνο μάλλον είναι κομμάτι τη συνολική συμφωνία επανεισδοχή επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Τουρκία. Τώρα για τι ομάδε, τι ευρωπαϊκέ ομάδε ε, συνοριακών φυλάκων. Δύο βασικοί στόχοι. Πρώτο βασικό στόχο είναι να χρησιμοποιήσουμε μια υφιστάμενη δεξαμενή τέτοιων υπαλλήλων. Τα κράτη-μέλη ήδη αναπτύσσουν αξιωματούχους επισκέπτες guest officers έξω από αυτές τις δεξαμένες. Εμείς θέλουμε εμπειρογνώμονες που δίνονται σε αυτές τις δεξαμενές, σε αυτά τα πουλ, ώστε να έχουμε τα άτομα που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση που χρειαζόμαστε. Και αυτός είναι και από τους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούμε στον Frontex. Να χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έπειτα, για τον αριθμό των εμπειρογνώμων. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου χίλιους εμπειρογνώμονες στη δεξαμενή. Τι κάναμε πρόσφατα να ξαναδούμε το προφίλ όλων των πυρογνωμόνων και να διευκρινίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση βάσει των διατάξεων του κανονισμού. Ο στόχο μα λοιπόν είναι να ξεκαθίσουμε καλύτερα αυτή τη δεξαμενή. Να απαντήσω τώρα στην κυρία Ρομέρο για την Ιγυρία. Είπατε πώ αποφασίζουμε με ποια χώρα ξεκινούμε τι Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Προκύπτει ο λόγος από την ανάλυση κινδύνου. Στην Ιγυρία είναι προφανές ε, το γιατί. Είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο που μας δίνει τους παράνομους μετανάστες και επίσης είναι μια χώρα πηγή ε, διακίνησης ανθρώπων. Άρα δικαιολογείται η επιλογή. Επίσης υπάρχει και μία συνάφεια με την ε, πολιτική ε, εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση των τρίτων χωρών να συνεργαστούν μαζί μας. Και αυτό είναι ένα από τα πλέον δύσκολα, ε, όπως φάνηκε στο παρελθόν. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες. Αλλά άμα δεν θέλει και η άλλη πλευρά, πώς θα γίνει. Με τη Σομαλία δεν έχουμε ακόμη μια τέτοια δυνατότητα, μια τέτοια πραγματικότητα για να προσεγγίσουμε Σομαλία. Προς το παρόν έχουμε 15 τέτοιες χώρες εταίρους, με τις οποίες έχουμε μια διευθέτηση εργασίας, έχουμε ανταλλαγές απόψεων, ε, προς, πληροφοριών, συγγνώμη, όχι προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο εκπαίδευσης, και κάποια εκπαίδευση που γίνεται μέσω των κοινών επιχειρήσεων. Είτε με παρακολούθηση, είτε με συγχρονισμό των κοινών επιχειρήσεων με τις χώρες. Στην περίπτωση της εστιάζουμε ιδιαίτερα στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφών. Ε, είναι η παριθμόν ένα χώρα για την οποία κάνουμε επιστροφές. Για το άσυλο, η πηγή μας είναι το δίκτυο ανάλυσης κινδύνου του οργανισμού. Δηλαδή, παίρνουν πληροφορίες για 8 δείκτες. Ένας εξ αυτών είναι ο αριθμός των ετούντων άσυλο υπάρχει η οργάνωση των ενδιαφερομένων μερών των κρατών μελών που μας δίνουν τα στοιχεία. Επίσης υπάρχουν στοιχεία από την Eurostat. Και η ΕΑΣΟ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου, θα έχει στο μέλλον και πιο αξιόπιστα στοιχεία, πιστεύω. Αλλά βασικά αυτά είναι στοιχεία αναφοράς. Και έτσι συγκρίνουμε τις τάσεις. Ο Frontex δεν συμμετέχει σε, δεν συμμετέχει, συγγνώμη, σε διαδικασία ασύλου. Το καθοριστικό σημείο είναι το screening που γίνεται. Δηλαδή, ο guest officer κρίνει αυτό το άτομο θα μπει σε δικασία ασύλου, οπότε δεν είναι θέμα ελέγχου συνόρων, είναι θέμα ασύλου. Και εκεί αποσύρεται. Για την κυρία Κέλλερ, για τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ελπίζω να απάντησα. Ήδη έχει ξεκινήσει η δικασία, χρειαζόμαστε όμως και την ε, δυνατότητα να πληρώσουμε αυτή τη θέση οικονομικά. Τα κριτήρια. Όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός, μπορούμε να αναστείλουμε, να αναβάλουμε και ποιος είναι τρίτος όρος, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, την κοινή επιχείρηση μπορούμε να την αναβάλουμε, οπότε τα κριτήρια υπάρχουν. Ρωτήσατε κάτι για τη ΣΥΠΑ. Ναι, το 18% των αρνήσεων εισόδου που αποφασίζουν οι Βρετανικές αρχές αφορούν Αμερικανούς υπηκόους. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι σπουδαστές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια. Δεν έχουν όλα τους τα έγγραφα και αυτή τη στιγμή τα έγγραφα δεν αρκούν, άρνηση εισόδου. Είναι μια σταθερή τάση που φαίνεται. Πολύ ψηλός ο αριθμός υπηκών νομένων πολιτιών που την χάνουν άρνηση εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την Λιβύη που ρώτησε ο κύριος Κροτσέτα, που είμαστε στο... αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το πρόγραμμα για την αύξηση του δυναμικού, το capacity building ε, στη Λιβύη. Και όταν οριμάσουν συνθήκες, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι τις προσπάθειες συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Κομισιόν δουλεύουν αυτό το σχέδιο, το capacity building, και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη δικασία σε ό,τι αφορά την έρευνα και διάσωση. Κάθε θαλάσσια επιχείρηση έχει ως σκοπό να κάνει ό,τι είναι δυνατό και εφικτό να σωθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ο Frontex όμως δεν ηγείται αυτών των επιχειρήσεων. Το βασικό σύστημα βάσης των μάλλον αυτό που ουσιαστικά θέτει να αμφιβόλω την αποτελεσματικότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι ε, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσιδιάσωσης ε, και δεν είναι πάντοτε το ίδιο κέντρο που αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο στο συντονισμό αυτών των επιχειρήσεων διάσωσης. αν ε, υπάρχει πρόβλημα με ανθρώπους, τότε αποστέλλεται σχετική έκθεση στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διεύθυνση Θάλασσα και εκεί αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο ο πλέον αρμόδιος. Και φυσικά διαβιβάζεται η αρμοδιότητα συνεχώς. Και κάποιες περιπτώσεις υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των σχετικών αρχών των κρατών μελών. Επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν συμμετέχουμε άμεσα στην διαχείριση ε, και στην αλυσίδα ε, εντολής. Ελπίζω ότι απάντησα στις περισσότερες τουλάχιστον ερωτήσεις. Α, ETPS, με ρωτάτε. Α, αυτή την ερώτηση κάνατε και δεν μπόρεσα να την κατανοήσω καλά. Δεν μπήκα σε όλες τις λεπτομέρειες, γι' αυτό. Για την ε, αρχή προστασίας δεδομένων. Αλλά και εμείς εργαζόμαστε επ' αυτού, αλλά και σε στενή συνεργασία με την αρχή προστασίας ε, δεδομένων και με τους άλλους οργανισμούς, σύμφωνα με τους ε, τεθειμένους κανόνες. Αλλά μόλις θα έχω περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορέσω να σας πω. Μία ωστόσο άλλη ερώτηση που δεν απάντησα είναι του κ. Μπουσούτιλ σχετικά με τα δύο κριτήρια, το υποχρεωτικό και το δυνητικό, το must και το may του κανονισμού του Frontex. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τις προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε με τα must και τα may πέφτουν πιο κάτω στη λίστα προτεραιοτήτων. Από την άλλη μεριά, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πράγμα του νέου κανονισμού, που να περιέχει τον νέο κανονισμό δηλαδή, και που να μην έχουμε αρχίσει να μελετούμε την εφαρμογή του. Μπορεί να προχωρήσει βέβαια σε άλλο έτος μέσα στο πολιετή αυτοσχεδιασμό, 13, 14, 15 και ούτω καθεξής. Αλλά αν δεν μπορούμε να το κάνουμε φέτος, τότε θα πρέπει να το υλοποιήσουμε, θα έλεγα ίσως με κάποιο πιο μακρόπνο τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Κυρία Ρωμέρο Λόπες, μια σύντομη ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, μια και έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Δεν μου απαντήσατε σαν ερώτημα. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό των ε, λαθρέων ε, που δεν κρατούνται στα σύνορα και μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Πειράτεια. Αυτό αφορά τα χερσαία σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, τα εναέρια σύνορα μας ενδιαφέρει αυτό και δεν μου απαντήσατε. Και επίσης, όταν είπατε ότι η Νιγερία είναι η τέταρτη χώρα που δίνει ελευθερούς μετανάστες, ποιες είναι οι τρίτες πρώτες πριν από την Νιγηρία. Thank you. <coughs> please answer. Απαντήστε σας παρακαλώ. Ε, συγγνώμη που δεν ήμουν τόσο ακριβή στην απάντησή μου. Να λοιπόν τα νούμερα για το 2011 οι 141.000 απορρίψεις εισόδου και επιστροφές. Περιπτώσεις που ανακαλύφθηκαν. Ουδής γνωρίζει βέβαια τον πραγματικό αριθμό και αυτό είναι, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τις αστυνομικές δυνάμεις. Λοιπόν, 50 με 50% μεταξύ ε, χερσαίων και θαλάσσιων σύνορων. Προηγουμένως ήταν κυρίως τα ε, χερσαία σύνορα λόγω της Αραβικής Ανοίξεως τώρα είναι περισσότερο τα θαλάσσια, είναι μάλλον στα ίδια με τα θαλάσσια σύνορα. Οι σημαντικότερες εθνικότητες έχουν ως εξής, όπως τις βλέπετε, με τα νούμερα από την Αραβική Άνοιξη, όπως λέχθηκε τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αντιπροσωπεύουν 61 με 62 χιλιάδες περιπτώσεις, περίπου το ίδιο, δηλαδή το ίδιο αριθμό με την Κεντρική Μεσόγειο. Το ερώτημα είναι τι γίνεται, τι απογίνονται τα πρόσωπα αυτά. Αυτό είναι βέβαια το κέριο ερώτημα. Μετά από την κράτηση, μετά από την ανακάλυψή τους μάλλον, γίνεται σύλληψη. Μετά από τη σύλληψη συνήθως γίνεται μια καταγραφή, ένα screening και μετά οι εθνικές αρχές προσπαθούν να επεξεργαστούν τις περιπτώσεις αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να χωρίσουν τις περιπτώσεις ασύλου και τις επιστροφές. Υπάρχουν βέβαια πολλά βήματα που πρέπει να περάσει η, μια επιτυχημένη διαδικασία επιστροφής. Οι περισσότεροι πάντως που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος της επικράτειας επιστρέφουν εθελοντικά. Ο αριθμός που έδωσα είναι το μικρό ποσοστό όλων των διαδικασιών επιστροφής. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τις απαντήσεις. Θα πρέπει να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν η οποία επίσης έχει λάβει, έχει δεχθεί ερωτήσεις. Μια πολύ σύντομη απάντηση. Πολύ σύντομα, η Κομισιόν βέβαια επιθυμεί να εκπληρώσει τις νέες υποχρεώσεις που της ανατέθηκαν από τους νομοθέτες με την αναθεώρηση του κανονισμού Frontex και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο ενισχύσαμε την ομάδα μας των ανθρώπων που εξετάζουν τις επιστροφές, όχι μόνο τη Γενική Οδηγία Επιστροφών, αλλά εξετάζουμε και πιο προσεκτικά το τι γίνεται στις κοινέ επιχειρήσεις επιστροφής της Frontex. Άρχισε η εφαρμογή αυτή στα μέσα Δεκεμβρίου του 2011. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αφετηρία των δραστηριοτήτων αυτών. Η Κομισιόν θα προσπαθήσει να συλλέξει τις απαραίτητες εκθέσεις για να μπορεί να παρακολουθεί πολύ στενά όλες τις επιχειρήσεις που θα διεξαχθούν φέτος και βεβαίως θα αναφέρει στο Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται και από τον νέο κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονόματος των συναδέλφων, ιδίως τον κύριο Λάιτενεν για τις απαντήσεις του. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας φέτος. Εδώ λίγη η συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 9 Φεβρουαρίου και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.